So, liebe Kollegen. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Χαίρομαι που είστε όλοι εδώ. Τώρα όλοι τρόπος του λέγειν. Αναλογικό ήταν υπάρχουν προβλήματα με τις πτήσεις και εγώ δεν μπόρεσα να έρθω αεροπορικός, χρειάστηκε να έρθω με το τρένο, αλλά ανωτέρα βία δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό φυσικά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οδύνη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων και των οικείων τους. Αυτά που τραβάμε εμείς είναι ίσονο σημασία στα λεωφορεία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν στο πετσί τους τις συνέπειες ε, των τρομοκρατικών επιθέσεων. Γι' αυτό θα ήθελα στη μνήμη τους να κρατήσουμε ενός λεπτού Danke Σας ευχαριστώ. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη της συνεδριασής μας. Δεν ζήτησε κανείς τροποποίησή της, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνομαι την ημερήσια διάταξη. Σημείο πρώτο. Ανακοινώσει του Προέδρου. Στι 30 Μαρτίου έγινε η διάσκεψη κορυφη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση-Ινδία. Μία ακόμη διάσκεψη κορυφή. Ε, σημαντικό πολιτικό θέμα, γιατί από τον Απρίλιο του 2013 συζητάμε με την Ινδία την πιθανότητα σύναψη εμπορική συμφωνίας. Αλλά δυστυχώς δεν διαφαίνονται ακόμη πιθανότητες πρόοδου. Πάντως, ο διάλογος συνεχίζεται. Στις 17 Μαρτίου η Επιτροπή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις για τη βελτίωση των εμπορικών μας σχέσεων με την Τουρκία. Είχαμε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων και θέμα τον εξυγχρονισμό της Θελωνιακής Συμφωνίας με την Τουρκία. 29 Μαρτίου πάνελ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου με θέμα τη μέθοδο προσαρμογής του κόστους σε περίπτωση διαδικασίας αντι-dumping, κυρίως για τα, το βιολογικό ντίζελ από την Αργεντινή. Τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα, μέτρια. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, υποβάλει διεξοδικά τη διαδικασία αυτή και να μας ενημερώσει για τις αποφάσεις αυτού του πάνελ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Εμείς θα παρακολουθούμε πάντως εξελίξει στο θέμα αυτό. Γιατί δεν έχουμε ακόμη θωρακίσει το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου, της βιωσιμότητας ή τις τον των κριτηρίων για το βιολογικό ντίζελ. Όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν. Και τελευταία ανακοίνωση. Στη γραμματεία έχουμε νέα υπάλληλο, Μαρή Καλόμπικα. Θα μας ενισχύσει στη γραμματεία. Καλώς ήρθατε και Ελπίζω να έχουμε αγαστή συνεργασία. Αυτά ως προς ανακοινώσεις. Σημείο 3 τώρα. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας 15ης και 16ης Φεβρουαρίου του 2016. Όπως πάντα, μέχρι το τέλος συνεδρίασης ε, δεν υποβάλλεται παρατηρήσει ή αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 4 μακροπιστωτική, μακροοικονομική συνδρομή προς την Τινησία. Όπως γνωρίζετε, υιοθετήσαμε μια συμφωνία 300 εκατομμυρίων ευρώ για το 2014, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Τινησία, ε, μετά την Αραβική Άνοιξη και τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν πολλές ε, σε πολλές αραβικές χώρες. Έχουμε λάβει και το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ξέρετε. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα της Τινησίας για να μπορέσει η χώρα αυτή να εξελιχθεί όσο πιο εύρυθμα γίνεται. Είναι απαραίτητη λοιπόν αυτή η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και μάλιστα ψηφίσαμε και τις δεσμολογικές προτιμήσεις για το ελαιόλαδο και την επέκταση της ποσόστοσης. Κυρία Ντεσαρνές, αν θυμάστε, ήταν η συγκεκριά μας. Έχουν απομείνει κάποιες εκκρεμότητες στη συζήτηση στο Συμβούλιο και τώρα επιλαμβανόμαστε θέμα της χορήγησης περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Τινησία. Θα ήθελα επευκαιρία να καλωσορίσω και τον πρέσβη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να του δώσω αμέσω το λόγο. Κύριε Σαρίφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισίας και ιδιαίτερα την ανάγκη μακροοικονομικής μικρής χρηματοδοτικής ε, συνδρομής προς την πατρίδα μου, δεδομένης της παρούσας ε, ε, πολιτικής κατάστασης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, για τα έκτακτα εμπορικά μέτρα που υπερψηφίσατε υπέρ της θυνησίας και την επέκταση της ποσότητας ελαιολάδου που εξάγεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η θετική ψήφος δείχνει τη δέσμευση και την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλευρό της θυνησίας σε αυτή την προσπάθεια δημοκρατικής μετάβασης που έχει ξεκινήσει το 2011 και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Θα συμφωνείτε ότι μέχρι στιγμής η Ισία έχει διανύσει πολύ δρόμο από το 2011 σε αυτή τη νέα δημοκρατική φάση που βρίσκεται. Βέβαια αυτή η αναδυόμενη δημοκρατική κατάσταση αντιμετωπίζει σήμερα μια έκτακτη, ασυνήθιστη κατάσταση τεράστιων προκλήσεων στο θέμα της ασφάλειας και με μια περιφερειακή συγκυρία δυσμενή εξαιτία τη κρίση στη Λιβύη αλλά και κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις, πολέμηση της ανεργίας που ανέρχεται σήμερα στο 15,4% με μεγάλο ποσοστό ανεργίας των νέων. Οπότε η απασχόληση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μείζονες προτεραιότητες. Και μάλιστα οι διαμαρτυρίες που έγιναν το, το 2016 σε πολλές πόλεις δείχνει την ανάγκη να εξασφαλίσουμε πιο εύρυθμη κοινωνικο-οικονομική μετάβαση. Για να αντιμετωπίσει προκλήσεις αυτές, η την υπολογεί σε μια έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μείζον ε, εταίρος της. Επίσης, 500 εκατομμύρια ευρώ ε, είναι επιπλέον ε, χρηματοοικονομική, μακροοικονομική συνδρομή που εξετάζουμε σήμερα. Εγώ θα είχα ζητήσει φυσικά πολύ περισσότερα από 500 εκατομμύρια, γιατί την Ισία, δεδομένης της κατάστασης, χρειάζεται 5 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 500 εκατομμύρια. Βέβαια, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα δάνειο 2,8 δισεκατομμύρια, γιατί όπως σας είπα η Τινησία χρειάζεται 5 δισεκατομμύρια. Και επιπλέον ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ε, θα ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα ένα επιπλέον δισεκατομμύριο. Γιατί η κατάσταση το απαιτεί. Πρόκειται για έκτακτο μέσο, έκτακτη συνδρομή για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές μας δυσκολίες, αλλά και να στηρίξουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε ξεκινήσει, προκειμένου να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια υφόρο ανάπτυξη που θα ωφελήσουν όλο τον πληθυσμό της Τινησίας. Και μάλιστα οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στο 2015 στην Τινησία ε, γονάτισαν την ίδια έθραυστη κατά την οικονομία μας. Και μάλιστα το 2014 είχαμε 2,3 ανάπτυξη και τώρα μόνο 0,8%. Και ο τουρισμός που είναι βασικός τομέας της οικονομίας με 7% του ΑΕΠ και 14% της απασχόλησης και 10% συνάλλαγμα έχει μειωθεί 35% το 2015 και 50% συρρυκνωθεί το 2016 εξαιτία τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο τουρισμός απασχολεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους άμεσα ή έμεσα. Οπότε, ήδη έχουμε 15,4% ανεργία, ε, με ένα πληθυσμό 11 εκατομμύρια, 15,4% του ενεργού πληθυσμού στην ανεργία, συν ένα εκατομμύριο οικογένειες που άμεσα ή έμεσα ζουν από τον τουρισμό, σκεφτείτε τι τεράστιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε λόγω της κατάστασης και στον τουρισμό και τη αυξημένη ανεργίας γενικώ. Άλλες ε, κινητήρες δυνάμεις οικονομίας επίσης ε, έχουν υποστεί επιβράδυνση. Μειώθηκαν οι εξαγωγέ εξαιτίας των κοινωνικών διαμαρτυριών, ιδιαίτερα στον τομέα των ορυχείων. 77% των εξαγωγών ε, της γίνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, κατάσταση στη Λιβύη. Πέμπτος οικονομικός μα εταίρο ήταν η Λιβύη πριν την κρίση. Αλλά και με τις αλλοδαπές επενδύσει είχαμε μια μείωση 5,6% την τελευταία πενταετία. Έτσι μειώθηκε η συμβολή του στι γενικέ στις γενικές επενδύσεις και στο ΑΕΠ. Και επηρέασαν κυρίω την απασχόληση αυτέ οι μειωμένε αλλοδαπέ επενδύσει. Γιατί για να δημιουργηθούν τι απασχόληση χρειάζονται επενδύσει πέραν αυτών των δυσχεριών της οικονομίας έχουμε και πρόβλημα με την ασφάλεια, κάτι που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Το 2016 πάνω από το 20% του προϋπολογισμού μας θα αφιερωθεί σε δαπάνες ασφάλειας και άμυνας. 30% επίσης μέχρι στιγμής αφιερώναμε στην παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό και τώρα ό,τι αφιερώνουμε στην παιδεία, ένα τμήμα θα το κατευθύνουμε σημαντικό στην άμυνα και την ασφάλεια. Αναφυσβήτητα, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία έχει τεράστιο οικονομικό και χρηματοοικονομικό κόστο. Ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη, το βάρο του είναι διαφορετικό. Πολλές λοιπόν οι προκλήσεις και γι' αυτό οι αρχές αποφάσισαν να κάνουν τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις για να ανακάμψει η οικονομία και ένα αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2016-2020 βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης. Έτσι φαίνονται οι προτεραιότητες της τινησιακής κυβέρνησης για να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο οικονομίας που θα εξασφαλίσει αηφόρο ανάπτυξη και ακριβωδίκη κατανομή των πόρων καθώς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης ένα εξαντλητικό πρόγραμμα κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνεται σε αυτό το νέο σχέδιο. Πέντε είναι οι άξονε των νέων μεταρρυθμίσεων. Χρηματοδότηση τη οικονομία πρώτο, ανάπτυξη των ισορροπιών των οικονομικών, πρόθεση του ανθρώπινου δυναμικού και των ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ενό δικτύου κοινωνική προστασία ε, με μεταρρύθμιση των κοινωνικών ταμείων ασφάλιση και αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου. Επ' θέλω να σας φέρω και το, το νέο νομοσχέδιο για την Κεντρική Τράπεζα της Τινησίας και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και ένα νέο παιδικό σχέδιο που ε, εξετάζεται αυτή τη στιγμή στην Ισιακή Βουλή. Δεδομένων των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και των ε, σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τη Τινησίας, ε, για φέτο έχουμε υπολογίσει την ανάγκη εξωτερική χρηματοδότηση στα 5 περίπου δισεκατομμύρια. Η πρόθεση μακροοικονομικής ε, χρηματοδοτικής συνδρομή 500 εκατομμυρίων θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε εν μέρη τις ανάγκες μας ε, με ε, ευνοϊκό επιτόκιο, μακρο, μέσο πρόθεσμα, ώστε να μην χρειαστεί να αποταθούμε στις διεθνείς αγορές με υψηλά επιτόκια. Επίσης, θα βελτιώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις δημοσιονομικές μας και κυρίως θα στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θέλουμε να ενισχύσουμε την αηφόρα μας οικονομία και την ανάπτυξή μας. Λυπάμαι που μακρηγόρησα. συνήθω δεν μου αρέσει να διαβάζω τι ομιλίε μου. Αλλά οι συνάδελφοι μου πρέπει αυτά να τα διαβάζουμε, να τα γράφουμε και να τα διαβάζουμε για να μην ξεχάσουμε τίποτα. Και μετά την πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή του 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο, κυρίως αναθεωρώντας προς τα πάνω τα δάνεια που δόθηκαν προς την Τινησία. Ήταν σημαντική λοιπόν η αρρωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσβλέπουμε και στη νέα υποστήριξη για τη νέα αυτή συνδρομή. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα συμπληρωματική χρηματοδοτική συνδρομή, το συντομότερο δυνατό, στην πρώτη εκταμείευση να γίνει δυνατό και πριν το καλοκαίρι. Οι τινησιακέ αρχέ ε, έχουν δεσμευτεί να επιταχύνουν τι σχετικέ διαδικασίε. Και θα ήθελα εγκατακλείδη να επαναλάβω την ευχή μου να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίζει τις προσπάθειες υπέρ της δημοκρασίας της που είναι πολύ ευάλωτες και να συνεχίσει τον εκδημοκρατισμό της και την οικονομική της σταθεροποίηση. Και σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Je, je, je remercie beaucoup. Κυρία ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον κύριο Πρέσβη, ο οποίο, όπω ε, πάντα μα περιέγραψε την κατάσταση στην ε, χώρα του και τα έχουμε πει διαμακρών για όλα αυτά τα ε, κείμενα και μιλήσαμε για αυτή την ε, εξαιρετική εξαιρετικού ρύθμιση που αφορά τι ποσοστώσει του ελαιολάδου. Όπω μα τα είπε ο κύριο Πρέσβη, όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Τινησία. Ε, είναι πάρα πολύ λεπτικέ οι ώρε, οι δύσκολε, η συγκυρία. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα και προκλήσει που αντιμετωπίζει και θα πρέπει να αντιδράσει κανείς για όλα αυτά τα προβλήματα και είναι και το θέμα της ασφάλειας όπως είπε ο κύριος Πρέσβης κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων ε, γιατί πρόσφατα η Τινησία έπεσε θύμα τέτοιων επιθέσεων, άρα επομένω το διαγύβημα είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει σημαντική ανεργία, υπάρχουν πολλές ε, ανισότητες ε, στη χώρα. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της ανεργίας των νέων που αγγίζει το 40% ε, και ακριβώς πρόκειται για αυτές τις ανισότητες που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Όπως μας είπατε κύριε Πρέσβη, είναι τρομερό αυτό και είπατε για το 30% του προϋπολογισμού που πάει εις ε, την ε, παιδεία, οπότε και σήμερα αυτές, αυτά τα χρήματα πάνε τώρα σε άμυνα και ασφάλεια. Βλέπουμε επομένω το πόσο χρειάζεται την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα και όπως είπατε μιλάμε για 5 δισεκατομμύρια χρηματοδοτικές ανάγκες εμείς ε, πρόκειται ε, να βοηθήσουμε με 500 εκατομμύρια μακροοικονομική βοήθεια θα ακούσουμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε λίγο και θα ε, συναντηθούμε και πάλι για να δούμε πώς από τεχνοκρατικής πλευράς αυτά θα ρυθμιστούν οπότε συμφωνούμε με τους στόχους σας κύριε Πρέσβη, άρα θα πρέπει να γίνει εκταμείευση των πόρων το συντομότερο δυνατόν, πάμε για το καλοκαίρι και έτσι να πετύχουμε τη συμφωνία μεταξύ των τριών δεσμικών οργάνων ε, και έτσι θα πρέπει να ε, επιτελέσουμε το νομοθετικό μας έργο το συντομότερο δυνατόν. Αυτά κύριε Πρόεδρε προς το παρόν. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Λάγκε. Σας παρακαλώ τώρα, κυρία Σαφή. Σαϊφή, με συγχωρείτε. Με ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Πρώτα, μεταφέρω τις συγγνώμε του κυρίου Τσιπού που είναι, κολλείται σήμερα και βεβαίω αυτό οφείλεται και ενδεχομένω και σε κάποια προβλήματα μεταφορών που έχουν διαπιστώσει και άλλοι συναδελφοί μου. Ήθελα να πω και Πρέσβη, έως ε, πολλά έχουν ήδη και τα λέμε εδώ και μήνες. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε, δηλαδή πόσο πολύ σας υποστηρίζουμε και εσάς και τη χώρα σας. Και θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο με πολύ συγκεκριμένες δράσεις πέραν των λόγων και η ε, ε, συζήτηση αυτή για την μακροοικονομική στήριξη είναι πολύ σημαντική. Ε, πέντε χρόνια μετά από εκείνη την περίφημη Αραβική Άνοιξη, δεν θα σχολιάσω περισσότερο, η Τινησία είναι η μόνη χώρα που εξακολουθεί να ε, βρίσκεται σε μια δημοκρατική πορεία. Βεβαίως και ορισμένοι πολίτες έχουν λάβει και το βραβείο Νομπέλ. Και βέβαια η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι μια υπόθεση που χρειάζεται πολύ χρόνο για να γίνει σε βάθος και να έχει διάρκεια. Και είναι μόνο μια διαδικασία πολύ μακρά. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ποιες είναι οι προκλήσεις που συνδέονται με την ε, προσπάθεια αυτή και που ενδεχομένως την υπονομεύουν και την ε, θέτουν σε κίνδυνο. Αφενός η τρομοκρατία Αρχίσαμε την συνεδρίασή μας σήμερα με ενός λεπτού σιγή ε, στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων δύο βήματα από εδώ, στις Βρυξέλλες και πριν από λίγες μέρες πάλι άλλη επίθεση στην ε, την Ισία και αλλού στον κόσμο. Όλοι πληττόμεθα από την μάστιγα αυτή. Επίσης οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Θυμάμαι η πρώτη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου που είχε μεταβεί στην Τινησία Μαριέλ μαζί σας αμέσως μετά την εξέγερση αυτή. Ήδη δημιουργούνταν πολλά κοινωνικά κινήματα διότι για του τους ε, πολίτες δημοκρατία σημαίνει βελτίωση άμεσα της κοινωνικής τους καταστάσεως. Βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί η Τινησία σε όλες αυτές τις σημαντικές προκλήσεις. Και βεβαίω ε, μίλησα και για τι επιθέσει που λαμβάνουν χώρα δυστυχώ τακτικά. Ο νησιακό λαό και οι εκπροσωποί του θα πρέπει να δείξουν επιμονή, ε, φιλοδοξία για του στόχου τη πατρίδα του. Και είμαστε στο πλευρό σα. Αυτή λοιπόν η μακροοικονομική υποστήριξη για την, την είναι σημαντική. Αναπτύξατε επιχειρηματά σα κύριε Πρέσβη. Είπατε ότι μάλλον χρειάζονται 5 δισεκατομμύρια είναι τεράστιες οι ανάγκες σας βεβαίως. Είναι σημαντικό πάντως εμείς ήδη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό και μάλιστα γρήγορα. Θέσατε επίσης ένα θέμα που γνωρίζουμε όλοι και που είναι η ανεργία των νέων. Άλλη μάστιγα αυτή, μεγάλη πρόκληση και η οποία μάλιστα πλήττει και τις δυο πλευρές της Μεσογείου γνωρίζουμε και εμείς το πρόβλημα αυτό. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα από τα λόγια στις συγκεκριμένες πράξεις και ας σταθούμε στο πλευρό του λαού σας, της Τινησίας και του Τινησιακού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η κυρία Δεσάρνες και η κυρία Σαϊφή ήταν σαφέστατε, στο ίδιο και ο πρέσβης της Τινησίας. Η Τινησία αντιμετωπίζει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Ε, γίνεται πολλούς λόγους για την Αραβική Άνοιξη. Μάλιστα, εγώ ε, είχα μιλήσει με τον κύριο Χαϊσέψη, τον ε, σημερινό πρόεδρο της Τινησίας, όταν ήταν απλώς ε, πρόεδρος του κόμματός του. Είχα λοιπόν ε, μιλήσει μαζί του και του είχα πει η Αραβική Άνοιξη και μου είπε όχι, Μην λέτε Αραβική Άνοιξη, να λέτε καλύτερα Αραβικός χειμώνας ίσως λοιπόν αυτή η άνοιξη είχε κάποια αρνητικά τελικά αποτελέσματα και κάποιους αρνητικούς καρπούς. Πάντως η Τινησία είναι ένα υπόδειγμα. Είναι η μοναδική αραβική χώρα που έχει πραγματικά μια δημοκρατία αυθεντική ε, κατά τα δυτικά πρότυπα. Και είναι ένα κακό παράδειγμα για τον ΤΑΕΣ. Γι' αυτό θα προσπαθήσει τον ΤΑΕΣ να υπονομεύσει αυτήν την ε, δημοκρατία στη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε με κάθε προσπάθεια την Τινησία και με οικονομικές προσπάθειες ε, να έχουμε ένα είδος σχεδίου Μάρσαλ για την Τινησία που είναι μικρή χώρα και χρειάζεται να καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Επίσης είναι σημαντικό στην Αθηνά και χείρακη είναι, δηλαδή και η νησία να έχει σταθερή κυβέρνηση, πιο συμπαγή, πιο συσπηρωμένη, με λιγότερες διχόνε και διαιρέσει. Το θέμα της ασφάλειας φυσικά έχει ζωτική σημασία, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν θα έχει τουρισμό και ούτε ευρωπαϊκέ επενδύσει η χώρα αυτή. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη η παράκτητη νησία και η την νησία των μεγάλων πόλων δεν έχει καμία σχέση με την ενδοχώρα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και όσο συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας, ε, δεν θα έχουμε σημαντική πρόοδο. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως στην ενδοχώρα της νησίας Και ας μην ξεχνούμε ότι η νησία είναι η δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό πολιτών κατά κεφαλήν ε, στο Ισλαμικό κράτος, ε, με τη, ως ξένοι μαχητές δηλαδή. Οπότε η Τινησία είναι η δεύτερη χώρα. Ε, είναι σημαντικό αυτό να το λάβει υπόψη την Ισιακή κυβέρνηση και να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο με κάθε προσπάθεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, αναφέρθηκε η κρίση στη Λιβύη, η καταβαράθρωση του τουρισμού, οι οικονομικές δυσλειτουργίες και δυσκολίες. Γι' αυτό και θα πρέπει ανεπιφύλακτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει και να συνδράμει την Τινησία, αλλά θα πρέπει και η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα που χρειάζονται αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ευχαριστώ. Ο, ο πρόεδρος, ευχαριστώ. David Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την πρόταση ο Εμμανουέλ Μορέλ. Είναι ο εκπρόσωπός μας για το θέμα αυτό, αλλά είναι απόν σήμερα δεν έχουμε καμία ψευδέστηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει την Ισία και όλοι οι μεγάλοι Βρετανοί tour operators, το βλέπω αυτό στις ιστοσελίδες τους, έχουν ακυρώσει τα ταξίδια προς την Τινησία φέτος. Όπως λέει ο πρέσβης, για μια χώρα που εξαρτάται τόσο από τον τουρισμό, αυτό είναι βαρύ το πλήγμα. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι ζωτική σημασία δοθήσεις της θέσεως της Τινησίας και απέναντι στον ΤΑΕΣ να στηρίξουμε την, την Ισιακή Δημοκρατία με κάθε δυνατό μέσο. Ευχαρίστω λοιπόν η πολιτική μου ομάδα στηρίζει τα αυτόνομα ε, μέτρα και τα 500 εκατομμύρια για την στήριξη. Δεν είναι ασήμαντο το ποσό, είναι βέβαια μικρό απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ε, την Ισία. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαθέσει όντως το 1 δισεκατομμύριο το οποίο έχει δεσμευτεί να διαθέσει. Και επίσης στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την σε βάθος εμπορική συμφωνία. Δεν θα λύσει αυτή τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα της Τινησίας, θα δώσει όμως μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη χώρα αυτή. Στηρίζουμε λοιπόν και την πρόταση αυτή και ελπίζω τα βήματα που θα ακολουθήσουν να είναι ταχύτατα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Λάγκε. Εσείς, Χέλμουτ Σόλτ. Στα αγγλικά. Και ο δικός μας και ο είναι απόν σήμερα. Μου ζήτησε να μεταφέρω ορισμένα, ορισμένες του προβλήματος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Αραβική Άνοιξη έχει επιφέρει ε, κάποιες δυσκολίες στην, και στην χώρα αυτή και όλους μας απασχολούν και πρέπει να δούμε ποια είναι τα ενδεχόμενα βήματα που μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουμε τους πολίτες της χώρας αυτής. Μιλούμε για μαζική ανεργία, ιδίω των νέων, Πώς μπορούμε άραγε να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων για να αποφευθούν παραπέρα προβλήματα και εντονότερα προβλήματα. Εδώ η μακροοικονομική υποστήριξη νομίζω μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που αυξάνει μέσω και μακροπρόθεσμα την χρέωση της χώρας, το χρέος της χώρας. Η ερώτηση λοιπόν είναι, χρειαζόμαστε όντως ως εργαλείο την μακροοικονομική υποστήριξη η οποία ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να επιβαρύνει, να δυσχεράνει την θέση της Τινησίας. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον κύριο Πρέσβη, τον οποίο ευχαριστώ για την ανάπτυξη των απόψεών του, είναι η εξής. Πώς κρίνεται την δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλο το φάσμα δυνατοτήτων που έχει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ε, οικονομίας της ε, την Ισίας. Ελαφρύνοντας το χρέος της Τινησίας μέσα από μια προσπάθεια να ανακτηθούν τα όσα έχουν ε, καταχραστεί οι διάφορες ε, ελίτ, οι προηγούμενες δηλαδή κυβερνήσεις και άλλες ελίτ της Τινησίας. Νομίζω πάντως ότι ε, η πολιτική υποστήριξη προς την Τινησία με ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ του δημοκρατικού κινήματος ε, της Τινησίας πρέπει οπωσδήποτε και αυτά να σταλούν και βεβαίως να προαχθεί και η οικονομική και εμπορική συνεργασία με, τα, με την, την Ισία. Μάλιστα, εσείς τώρα εκ των Πρασίνων, μάλιστα, σύντομη παρατήρηση, ο κύριος Μπούχνερ. Σύμφωνο με τα όσα λέχθηκαν και ιδίω σχετικά με τα προβλήματα που υπέμνησε ο κύριος Σόλτς. Νομίζω πάντως ότι και πέραν της Τινησίας έχει κέρια σημασία για μας οι εξελίξεις να κινηθούν προς την κατεύθυνση περισσότερης δημοκρατίας. Είπατε και εσείς ότι η Τινησία είναι η μοναδική χώρα που εγείρει κάποιες ελπίδες και που ελπίζω ότι θα μπορέσει έτσι να επηρεάσει και άλλες χώρες. Πάντως εμείς πρέπει να πράξουμε πάντα δυνατόν εδώ για την στήριξη της Τινησιακής Δημοκρατίας. Θα συμφωνήσω με τον Σόλτς και θα ζητήσω λιγότερο δάνεια, λιγότερα δάνεια, περισσότερο όμως μια και μακροπρόθεσμη στήριξη της χώρας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ecofinance, ποιος άραγε ε, την εκπροσωπή, εσείς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ξέρετε, η Τινησία είναι σε μια πολύ δύσκολη μακροοικονομική κατάσταση από το 2011 εξαιτία μια σειρά παραγόντων και συμπεριλαμβανομένων και των ε, εσωτερικών αναταραχών κατά την πρώτη φάση της πολιτικής μετάβασης, αλλά κυρίως εξαιτία της περιφερειακής αστάθειας. Η κρίση στη Λιβύη ε, αντικατοπτρίζεται αρνητικά και στην Τινησία, αλλά και εξαιτία ε, ε, της κατάστασης της οικονομικής και των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί η χώρα είναι ε, αυτή που ε, έχει 70% εμπόριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και τις περισσότερες εμπορικές συναλλαγές. Οπότε σε αυτήν την άποψη συμφωνήθηκε ένα πρόγραμμα στήριξης το 2013 με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που συμπληρώθηκε μετά το αίτημα για την πρώτη δόση 300 εκατομμυρίων ευρώ μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκτοτε εφαρμόζουμε αυτή τη συνδρομή. Ήδη έχουμε εκταμιεύσει δύο δόσεις από τα 300 εκατομμύρια, το Μάιο και το Δεκέμβριο του 2015. Έκτοτε όμως είχαμε νέες εξελίξεις, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας, ε, η χώρα έχει υποστεί πολλέ τρομοκρατικέ επιθέσει με ολέθριο αποτέλεσμα σε πολλού κλάδου τη οικονομία, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, με μείωση του τουρισμού πέρυσι κατά 40 με 45% ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού. Και τα τελευταία, τα πρόσφατα στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Για ε, το πρώτο τριμήνο του τρέχοντος έτους έχουμε ε, πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της του 50-55% του τουρισμού. Επιπλέον, η χώρα αντιμετωπίζεται, επηρεάζεται αρνητικά από μια δύσκολη κοινωνική κοινωνική κατάσταση. Είχαμε πολλές διαμαρτυρίες ε, από εργάτες στα ορυχεία κυρίως, ε, κάτι που ε, επηρεάζει την παραγωγή φωσφατούχων ουσιών και λιπασμάτων. Και η εσοδιά ήταν κακή εξαιτίας μιας ε, παραταμένης ανομαυρίας και μιας ε, συγκυριακής διόρθωσης εξαιτίας της περσινής κατάστασης του ελαιολάδου. Και η ε, γετνίαση με τη Λιβύα απαιτεί ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών και άρα ενισχυμένο προσωπικό ασφαλείας και στρατιωτικό προσωπικό. Εξού και το νέο αίτημα για περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα συνδρομή 500 εκατομμύριων ευρώ. Συνολικά βέβαια έχουμε 800 εκατομμύρια. Έχουμε ακόμη την τρίτη δόση που δεν έχουμε εκταμίευση από το, πρώτο το, το, το κομμάτι των 300 εκατομμύριων και τα 800 εκατομμύρια είναι από τα μεγαλύτερα ποσά χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ποτέ έχουν εκχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είπε η κυρία Δεσσαρνές, περιμένουμε τα 250 εκατομμύρια την πρώτη δόση της εκταμίευσης και δύο επιπλέον δόσεις από 100 εκατομμύρια. Θα θέλαμε να καταφέρουμε ήδη από τα τέλη του μήνα να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές του προγράμματος και αν όλα βγουν καλώς και συμφωνήσουν και τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής να εγκριθεί η πρόταση για τη χρηματοδοτική συνδρομή με σχετικά συνοπτική διαδικασία, αναμένουμε να υιοθετηθεί ε, η πρόταση ήδη από το Μάιο, ώστε να προλάβουμε να έχουμε την πρώτη εκταμίευση τον Ιούλιο. Γιατί η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή και είναι επίγοντο θέμα θα πρέπει η εκταμείευση να επισπευστεί στο έπακρο. Επίσης θα ήθελα να τονίσουμε και προς τον πρέσβη και προς τις ε, τρησιακές αρχές ε, την ανάγκη να διεκπαιρεωθούν οι συμφωνίες και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το συντομότερο δυνατό. Από τη στιγμή που θα λάβουν ε, τις νομοθετικές αποφάσεις οι αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνει συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές για την κύρωση του εγγράφου το συντομότερο δυνατό και από την Τινησιακή Βουλή, θα έχουμε το σχέδιο ώστε να μπορέσουμε την πρώτη δόση να την εκταμιεύσουμε πριν το καλοκαίρι και τη δεύτερη δόση κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η πρώτη δόση είναι 200 εκατομμύρια και οι επόμενες δύο από 150 εκατομμύρια. Το είχα κάνει λάθος στην αρχή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τωρινή είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ήδη εκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από το 2013 ε, μαζί με τις ε, κοινέ δηλώσεις με βάση τους κανόνες για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Έγιναν κάποιες ανεπαίσθητες τεχνικές αλλαγές ε, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και διευκρινίζοντας κάποιες διατάξεις ώστε να συνάδουν την κοινή δήλωση και τις προηγούμενες αποφάσεις. Ενθαρρύνουμε λοιπόν και καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό ε, στην έγκριση αυτή τη απόφαση. Το Συμβούλιο ήδη έχει ξεκινήσει τις συζητήσει και θεωρούμε ότι και το Συμβούλιο συμμερίζεται την ανάγκη και την, το κατεπήγοντα χαρακτήρα αυτής της απόφασης ώστε να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ω Κοινοβούλιο θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μα με ιδιαίτερη προσοχή ασφαλώς ως εκλεγμένο ε, σώμα ε, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ακούσουμε την εισηγήτριά μας, ή προτιμάτε πρώτα να ακούσουμε τον πρέσβη. Μετά εσείς πολύ καλά. Εσείς κύριε πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η 18η Απριλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα αρχίσει την Τίνιδα ο πρώτος γύρος και θα, ταυτόχρονα θα γίνεται και συνεδρίαση με συμμετοχή του ε, Υπουργού μου των Εξωτερικών και της κυρίας Μογκερίνη στο Λουξεμβούργο. Υπάρχουν πολλέ προσδοκίες από την Τινησία σχετικά με την ε, ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τινησία. Και πολλοί ακούν για ελεύθερε συναλλαγές. Εγώ προτιμώ μια συμφωνία στήριξης. Γιατί αυτό καθησυχάζει περισσότερο. Γιατί πολλοί επικρίνουν την συμφωνία αυτή στην την Ισία. Και για τη συμφωνία από το 1995 για τον βιομηχανικό τομέα και τη σχετική αξιολόγηση, η οποία αξιολόγηση δεν έγινε. Και πολλοί μιλούν για απολεσθέντα έσοδα του δημοσίου, του τιμησιακού δημοσίου δηλαδή, από την ιστορία αυτή. Και αυτή η εντύπωση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μιλούμε ε, συχνά για trade, not aid. Εγώ λέω trade και aid. Χρειαζόμαστε και τα δυο σε αυτού του είδους τις συμφωνίες, διότι μιλούμε σήμερα για μακροοικονομική συνδρομή, αλλά δεν πρόκειται για συνδρομή, δεν είναι δηλαδή βοήθεια. Είναι δάνειο με ευνοικού όρου, σύμφωνοι, αλλά παραμένει δάνειο, το οποίο οφείλει να επιστραφεί σε κάποια χρόνια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η χρέωση της ε, Τινησία βαρύνεται. Είχαμε πριν από την εξέγερση 44%, τώρα έχουμε φτάσει στο 53%. Ε, είναι διαχειρίσιμο το χρέο αυτό και ε, λογικό στο μακροοικονομικό επίπεδο. Όμως η κυβέρνηση έχει βάλει ένα 60% του ΑΕΠ που επιθυμεί να μην το υπερβεί. Φαίνεται η αύξηση να είναι τη τάξη του 5%, ήταν παλιά τη τάξη η ανάπτυξη τη Τάξη του 5%, τώρα έχουμε φτάσει στο 0,7% ή πάντως ένα μικρό ποσοστό. Ελπίζουμε να υπάρξει ξανά ανάκαμψη εάν είναι ευνοϊκέ οι συνθήκες, εάν βελτιωθεί το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν ξαναρχίζουν οι επενδύσεις. Είτε ενδοτινησιακές είτε και έξωθεν. Διότι η κατάσταση των επενδύσεων είναι ήδη αρκετά έθραστη σε όλο το Μαγκρέπ. Κανένα δεν πάει να περάσει διακοπέ του στην Τινησία ή να επενδύσει. Εκεί βρίσκεται η δυσκολία. Έχουμε περάσει και θετικές εμπειρίες και με συνεργασία με τη Γερμανία, με τη Γαλλία ε, με την μετατροπή ενός τμήματος του χρέους με τη Γερμανία αυτό αφορούσε 60 εκατομμύρια ευρώ, με τη Γαλλία το ίδιο και διοχετεύτηκαν τα χρήματα αυτά σε έργα αναπτυξιακά. Με τη Γερμανία το γνωρίζω διότι πριν ήμουν διευθυντής του τμήματος διμερών συμφωνιών. Έργα για το νερό, πόσιμο νερό στην αρχή και μετά ε, ε, βιολογικού καθορισμού. Αυτά τα πράγματα δίνουν ωστόσο ελπίδα, δίνουν, προσφέρουν απασχόληση, είναι καλά πράγματα. Τέτοια πράγματα θέλουμε να δούμε στην Τινησία. Να μας βοηθήσετε δηλαδή να δημιουργήσουμε πλούτο και επομένως ελπίδα για τους νέους. Αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμώ να περάσω σήμερα και σας ευχαριστώ και πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, η κυρία Σαρνέζ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αυτά που μας είπε ο κ. Πρέσβη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα πρώτα είναι σωστό να υπενθυμίζεται ότι ένα δάνειο αποκαλείται μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Όχι. Πρόκειται περί δανείου. Δανείου υπό όρους, υπό προϋποθέσεις περίπλοκες, δύσκολες, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση των δύο πραγμάτων και επομένω επ' αυτού έχετε δίκιο. και πάρα πολύ σωστά αυτά τα οποία είπατε, σαν παραδείγματα από Γαλλία και Γερμανία για αυτήν ε, την μετατροπή του χρέους και για την ε, μετατροπή του χρέους σε επένδυση. Οπότε είπαμε ότι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ζητηθεί το θέμα όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να δούμε ότι πάρα πολλέ δαπάνε στις χώρες είναι δαπάνε άμυνα και ασφάλεια που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία. Και η φύλαξη των ε, συνόρων αυτό τα, χιλιόμετρο χιλιόμετρα που την, από την Λιβύη, αυτό είναι θέμα Τινησίας αλλά και Ευρώπης. Και αυτό θα ήθελα να τονιστεί γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει την προβληματική μας για αυτή την κατάσταση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε από κοινού. Συνεργασία, αναβαθμένη συνεργασία, τεχνική, ε, πρακτική, ε, οικονομική και επίσης κάτι άλλο το οποίο μας είπατε είναι για το αλεκά και έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρει τα ίδια πράγματα. Το είπαμε ότι ίσως θα πρέπει να αλλάξει το όνομα και να μιλούμε περισσότερο, όχι για ελεύθερη συμφωνία ελευθέρων αλλαγών, αλλά για ε, μια εταιρική σχέση. Αλλά βέβαια θα πρέπει να αντιστοιχεί στον τίτλο και το περιεχόμενο. Η εταιρική σχέση αφορά την ανάπτυξη. Αλλά να, επί της ουσίας ποια είναι η διαφορά. Ανάπτυξη την Τινησία. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά τα οποία ε, εγκρίναμε ψηφίζοντας να ε, διακρίνονται από διαφάνεια και η σχετική συμφωνία να παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Δηλαδή, άλλα να συμφωνούμε και άλλα να κάνουμε. Να λαμβάνετε υπόψη ότι έχει συζητηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Άκουσα τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με αυτήν τη δέσμευση και όλοι θέλουμε να κάνουμε βήματα προόδου. Θα είπαμε ότι είμαστε οι νομοθέτες και έχετε προτείνει και αυτές τις ε, αποκαλούμενες τεχνικές ε, βελτιώσεις Άρα θα πρέπει να αναλυθούν αυτέ οι βελτιώσει. Επίση, θα πρέπει να δούμε και επί ουσία πώ το Συμβούλιο μπορεί να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί ε, όλα αυτά. Και θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα να εγκριθεί και να μην έχουμε καθυστερήσει. Και επομένω έτσι να δούμε πώ θα η πρόοδο στην υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Στα γερμανικά. Θα ξανασυζητηθεί, το σχέδιο εκθέσεως της κυρία Δεσαρνές στην συνεδρία της 21ης 22ης. Τώρα, θέμα υπαριθμών 5. Με την ένταξη της Κροατίας μεγάλωσε και η Τελωνιακή Ένωση. Και έχουμε τώρα βέβαια να συζητούμε με πολλές χώρες στα πλαίσια του ΠΟΕ. Μια από τις χώρες αυτές, δηλαδή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι η Κίνα. Και τίθεται τώρα επιτάπητο στο θέμα τη συμφωνίας μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα και ε, τη γνώμη μα συζητεί το Συμβούλιο, την οποία εκπονεί ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Βίγκλερ, ακριβώς όπως τονίσατε, συζητούμε για την διεύρυνση τη Τελωνικής Ένωση ε, μετά την ε, διεύρυνση προς την Κροατία. Οπότε αποφασίστηκε από το Συμβούλιο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ τα οποία άμεσα ε, καλύπτονται και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αντισταθμικές προσαρμογές σε περίπτωση που έχουν κάποιους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υψηλότεροι από τους αρχικούς ε, σχετιζόμενος με την Κροατία και σε διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΑΕ. Είδαμε ποιες θα είναι οι παραχωρήσεις και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. Έγινε ανταλλαγή επιστολών, υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας. Αυτά στις 7 Δεκάτου στις Βρυξέλλες και τώρα το Συμβούλιο αποφάσισε άρα επομένω θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία με αυτή την μορφή της ανταλλαγής των επιστολών. Έχουμε επίσης άλλους τέσσερις δασμούς για κάποια βιομηχανικά προϊόντα. Έχουμε μείωση δύο δασμών για ε, παπούτσια και κλιματιστικά και επίσης για το σκόρδο και για δύο είδη μανιτοριών. Κατά τη γνώμη μου είναι εύλογη η όρη αυτής της συμφωνίας και είναι προς συμφέρον μας να υποστηρίξουμε το ότι θα πρέπει ο Ευρωπαϊκή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στα πλαίσια του οργανισμού εμπορίου. Οπότε στα πλαίσια του σχεδίου ε, των προτασιών μας, πιστεύω θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτή τη συμφωνία. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο ουδή επιθυμεί να λάβει το λόγο. Τότε θα λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ομιλήσει. Κύριε Βίμπλερ, επιθυμείτε εσεί να δευτερολογήσετε. Τι να πω. Τι να πω, να βγάλω συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις και τα σχολεία μου. Ευχαριστώ πάντως όλε τις πολιτικές ομάδες για την υποστήριξή τους. φαίνεται ότι σημειώνεται ε, σημαντική συνένεση πάντως μεταξύ των μελών. Το υπαριθμόν 6. Η πρόοδος δηλαδή των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. δύο μάλιστα τριμερείς διάλογοι διεξάγονται με το Συμβούλιο. Κανονισμός κατά των βασανιστήριων και το άλλο είναι τα ορυκτά συγκρούσεων για την Anti-Torture Regulation. Θα θυμάστε πρόκειται για ήδη οι εμπορεύματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διεξαγωγή βασανιστήριων. Είχαμε δώσει με 600 ψήφους πλειοψηφία εντολή να διαπραγματευτεί η Επιτροπή εξ μας. Διεξήχθηκε δεύτερος τριμερής διάλογος όπου παρόλο που το Ευρωκοινοβούλιο είχε καταθέσει μια πραγματικά καλά θεμελιωμένη συμβαστική πρόταση, την οποία διαβίβασε μια εβδομάδα πριν από τον ημερή διάλογο η κυρία Σάκη στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε, δεν βρέθηκε σε θέση να διαβουλευτεί. Εμείς τονίσαμε ιδιαίτερα το θέμα που επιγράφεται στα αγγλικά ο sketch all, δηλαδή ο τελωνιακός υπάλληλος μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση όλων των εμπορευμάτων που μπορούν να παίξουν ρόλο σε βασανιστήρια. Αλλά χρειάζεται βέβαια και κανόνες για την διαμετακομιδή, το, το transit, δηλαδή την εμφάνισή τους σε εκθέσεις, την ε, διάθεσή του στο εμπόριο. Χρειάζεται λοιπόν και για όλα αυτά συγκεκριμένη εντολή, διαπραγματευτική εντολή. Δηλαδή, Δυστυχώ το Συμβούλιο, όπω είπα προηγουμένω, δεν αντέδρασε και δεν θεώρησε ότι είναι η θέση να διαπραγματευτεί. Όθεν αναμένουμε νέα θέση του Συμβουλίου. Η άλλη διαπραγμάτευση σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου που ε, διεξάγεται για τα ορυκτά συγκρούσεων πρώτος τριμερής διάλογος την 1η Φεβρουαρίου. Συναντηθήκαμε ξανά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Τρίτου, η οποία τροποποίησε την θέση της, ώστε αυτή να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με αυτήν του Κοινοβουλίου. Αύριο θα διεξαχθεί ο επόμενος τριμερής διάλογος. Και επ' αυτού να λάβει παρακαλώ ο κύριος Βίνκλερ ως εισηγητής μας τον λόγο. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα με μακρά ιστορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πολλά και διάφορα στοιχεία που είναι ελπιδοφόρα και ενθαρρυντικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρώσουμε αύριο. Δεν είναι και πολύ εύκολα τα θέματα, αλλά πολλά στοιχεία μας δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα στοιχεία και το Συμβούλιο περιμένει κάποια ανταπόκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, αύριο θα πρέπει να δώσουμε αυτά τα μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είμαστε πια σε θέση να λάβουμε απόφαση. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα μετά την Ολλανδική Προεδρία κατά το επίπεδο φιλοδοξίας του Συμβουλίου δεν θα παραμείνει τόσο υψηλό. Και μια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων θέλουν νομοθετικές διατάξεις για τα ορυκτά αυτά των συγκρούσεων, καλό θα ήταν να δώσουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να προχωρήσουμε και να δούμε και το θέμα του σχετισμού με την εξόριξη της έρευνας και την εξόριξη τέτοιων ορυκτών. Σήμερα και αύριο λοιπόν θα γίνουν συζητήσει και πιστεύω ω συζητητή ότι θα πρέπει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει το μήνυμα τη ελαστικότητα προ το Συμβούλιο και τη διαλλακτικότητα και τη ετοιμότητα να καταλήξουμε στη συμβαστική λύση με το Συμβούλιο με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επιτάπητο στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είναι ε, ταυτίζεται ακριβώς με τη δικιά μας, ε, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυμίες μας. Αλλά υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρία αυτή τη στιγμή που κράτησε δύο μήνες και πιστεύω ότι είναι όριμη η κατάσταση και προσφέρεται για συμφωνία με το Συμβούλιο. Υπάρχει γενικό σύμπνοια μεταξύ των μεγάλων πολιτικών, ε, σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων, οπότε θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόσφορο κλίμα. Επίσης, είναι σημαντικό να μην κολλήσουμε σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Τα αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για τα βασανιστήρια. Και φαίνεται ότι εκεί δεν θα προχωρήσει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Εκεί είναι πιο διάλακτη. Κάτι που δεν ισχύει για το θέμα για τα καύσιμα των συγκρούσεων. Ε, εδώ υπάρχει δυνατότητα πρόοδου. Πάντως διαπιστώνουμε ότι προετοιμαζόμαστε για την πολύ σημαντική συζήτηση για το θέμα της Κίνας που θα είναι και πολύ φλέγον και πολύ δύσκολο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην ε, έχουμε συσσωρεύσει και άλλα θέματα για να δούμε και το θέμα του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς για την Κίνα που θα είναι και πιο δύσκολο. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα με την σχετική νομοθεσία για το ρεκτά των συγκρούσεων και ευελπιστώ ότι αύριο θα έχουμε αμοιβαία σημάδια εμπιστοσύνη και μηνύματα εμπιστοσύνη από Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και ευελπιστώ και την πλουσία των πολιτικών ομάδων θα μας στηρίξει στο να καταλήξουμε σε έναν θετικό συμβιβασμό με το Συμβούλιο πολύ σημαντικό επαναλαμβάνω το θέμα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντικός εδώ. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα, για την έκβαση και πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε το ρόλο μας και στις τεχνικές διαδικασίες στη φάση της εφαρμογής αυτού του νομοθετικού οργάνου. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο και ειδικά η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, να εποπτεύσει τα πράγματα, ώστε κατά την προετοιμασία της εφαρμογής να μην αλλοιωθεί ή να μην αυληθεί το περιεχόμενο του κανονισμού. Και θα ήθελα να ξέρω και το δικό σας ρόλο, κύριε Πρόεδρε, στις διαπραγματεύσεις και από κοινού με τους και ηγητές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Πιστεύω ότι θα προσετεριστούμε το Συμβούλιο και θα το μετακινήσουμε κάπως προς τη δική μας κατεύθυνση. Θα ακολουθήσουν τεχνικές διαδικασίες, τεχνικοί διάλογοι. Πιστεύω ότι εκεί θα μας στηρίξει όσο γίνεται η γραμματεία. Ευχαριστώ, Ίνμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για αυτόν τον τριμερή διάλογο οποίος τώρα γίνεται σε σχέση με το ε, εμπόριο αυτών των αντικειμένων που σχέση με τα βασανιστήρια πάρα πολύ καλά μας τα εξήγησε ο Πρόεδρος, οπότε εγώ θα ήθελα να σας πω τα εξή δύο. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πούμε μπράβο στον εισηγητή για το έργο του. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να ε, μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις απόψεις όλων και βέβαια και στην τελευταία συνάντηση θα πάμε πάρα πολύ εισηγητικά όσον αφορά τις θέσεις του Συμβουλίου. Επίση, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι δεν μιλούμε για ακόμα μια ρύθμιση για εμπορία κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων. Μιλούμε για κάποια προϊόντα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο ή μπορεί να φορούν κάποιε τρομοκρατικέ επιθέσει που ακριβώ όλοι δυστυχώ έχουμε γίνει μάρτυρε τέτοιων, ε, τέτοιων, τέτοιων ενεργειών στη ζωή μα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια το Συμβούλιο και να φουγραστεί προσεκτικά τι λέει η Κομισιόν, τι λέει το Κοινοβούλιο που συμφωνεί μαζί μας και επομένως θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να κλείσουν αυτές τις συμφωνίες. Ε, θα πρέπει να σταματήσει αυτό το εμπόριο το οποίο στρέφεται κατά της ανθρώπινης ε, ζωής και επίσης θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη το ότι τα διοικητικά με τίποτα θα πρέπει φυσικά να κατησχύουν και να έχουν προτεραιότητα εναντί της ανθρώπινης ζωής. Άρα θα πρέπει επομένω να αναθεωρήσει το Συμβούλιο, να δείξει κάποια ευελιξία και να συντονιστεί με αυτό το πίστη το κοινοβόλιο. Χέλμουτ. Εγώ θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να επανήλθω ε, σε αυτά τα ορυκτά, τα επίμεχα. Και θέλω να θεωρήσω ότι έχει γίνει πάρα πολύ στη δουλειά και νομίζω ότι έχουν συνδυαστεί διάφορες ε, απόψεις ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχουμε μια καλή διαπαντευτική αφετηρία. Και επίσης θα πρέπει με κάθε ειλικρίνη να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όσον αφορά το θέμα τούτο και όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να δούμε το ότι τώρα ε, το περιεχόμενο προτάσεων μας είναι πάρα πολύ ποιοτικό, άρα θα πρέπει και το Συμβούλιο να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι προτίθενται να έχουν το μήκος κύματος μαζί μας και νομίζω ότι η ομάδα η διαπραγματευτική το πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ε, ε, σύμφωνοι στην γραμμή του και θα πρέπει εν ώψη των επόμενη συνάντησης να αποσπάσουμε κάτι συγκεκριμένο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με τι προτάσεις που έχουμε διαμορφώσει. Βέβαια να δούμε και τι θα πει το Συμβούλιο. Έχει το λόγο κύριε Φίζα. αυτά τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται και χρησιμοποιούνται τέλο πάντων για θανατική ποινή και για τα βασανιστήρια συμφωνούμε με, τον, με την συγκεκριμένη κυρία Σόλτ και νομίζουμε ότι ε, ε, έκανε δουλειά πάρα πάρα πολύ καλή γιατί το θέμα αυτό θα πρέπει να προωθεί στο Συμβούλιο δεν μιλάμε για οτιδήποτε ε, αντικείμενο για οτιδήποτε προϊόντα μιλάμε για κάποια προϊόντα όπω η κυρία Πινιέρη τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν για σοβαρέ παρεμβάσει των δικαιωμάτων. Άρα και εμεί θα πρέπει να είμαστε σκληροί στη γραμμή μα ε, και είμαστε ενωμένοι. Θα ήθελα πάντω να ακούσω τη γνώμη του Συμβουλίου. Νομίζω το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδείξει ευελιξία. Θα πρέπει να στηρίξει τι προτάσει του Κοινοβουλίου. Λέει ο κύριο Φίσα, πρόεδρο. Καλώς. Οπότε εμένουμε στις εξαιρετικές θέσεις μας και θα προσπαθήσουμε να τις προωθήσουμε. Θα σας κρατούμε ενήμερος πάντως. Σημείο 7. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων των ομάδων. Ουκρανία. 15 Μαρτίου έγινε η συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης ε, συνέχεια παρουσία του πρέσβη και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και εξετάστηκε η λειτουργία της Συμφωνίας Εμπορικής Σχέσης και Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία. Δυστυχώς δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια πρόοδο. Τώρα, τι θα γίνει ε, στις κατοχώρες, γιατί αναμένεται και το δημοψήφισμα για αυτή τη συμφωνία, τη σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία. Πολλά ερωτηματικά λοιπόν για το θέμα είναι μετέωρο και ελπίζω να μην χάσουμε εδώ τις κατοχώρες. Επίσης 15 Μαρτίου είχαμε την follow-up ομάδα για το Μερκοσούρ ε, με συμμετοχή των εμπορικών επιτετραμένων των πρεσβειών των χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Μερκοσούρ μάλλον. Εκεί διαπιστώνουμε κάποια ε, πρόοδο βέβαια και στην ε, Αργεντινή είχαμε κάποιες τροποποίησεις και στη θέση της Βραζιλίας. Αλλά μάλλον ε, θα περάσουμε σε εμβριθέστερες συζητήσεις. 16 Μαρτίου είχαμε την ομάδα ε, για την συμφωνία με την Τουρκία. δεν έχουμε καμία εξέλιξη εκεί. Επίσης 16 Μαρτίου η ομάδα για το follow-up για την Ιαπωνία. Ήταν και ο Μάριο Πετιτσίνη και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί διαπιστώσαμε μία νέα όθηση στις συζητήσεις. Αλλά αυτό το λόγο στο μόνιμο εισηγητή μα για το θέμα αυτό, τον κύριο Πέδρο Σίλβα. Ευχαριστώ. Συναντήθηκε στις 16 Απριλίου η ομάδα της παρακολούθησης με παρουσία του Μάριο Πετιτσάνη, του επικεφαλής των διαπραγματεύσεων που μας έκανε την ενημέρωση. Έχουμε νέα διαπραγματευτεί από πλευρά Ιαπωνία τον κύριο Ανεντά, που μας έδωσε κάποιες θετικές ενδείξεις ε, για ελπιδοφόρα εργαστή συνεργασία με τον νέο επικεφαλής ε, των διαπραγματεύσεων από πλευράς Ιαπωνίας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 15ο γύρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό σημάδι και από μόνο του. Οι Ιάπωνες μάλιστα κατέθεσαν και ένα κατάλογο με το 17% των προϊόντων που θα μπορούσε να ε, γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι το καλοκαίρι και ο επόμενος γύρος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και όλας στο Τόκιο. Παρ' όλα αυτά δεν αναμένεται ιδιαίτερη πρόοδος πριν το καλοκαίρι, γιατί θα γίνουν ε, εκλογές για την Άνω Βουλή της Ιαπωνίας. Η, η Ιαπωνία θέλει να εγκριθεί το TPP. Οι πιο ευαίσθητοι τομείς είναι η γεωργία και τα αγροεπιστητιστικά. Εκεί δεν περιμένουμε εντυπωσιακέ εξέλιξεις τις επόμενες εβδομάδες, το εγγύς δηλαδή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις θα εξελιχθούν σημαντικά μετά τις εκλογές αμέσως, μετά τις εκλογές, οπότε είναι ακόμη εφικτός ο στόχος του, 2016 για τη σύναψη της συμφωνίας, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αλλά πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο της διεκπαιρέωσης κατά το 2016. Άλλη ομάδα παρακολούθησης ε, συνεδρίασης της 17 Μαρτίου για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είχαμε εκτενή συζήτηση με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, τις υπηρεσίες και επιστήμονες και πυρογνώμονες. Η κυρία Ρένα δυστυχώς απουσιάζει σήμερα, κολλείται αλλά στην επόμενη συνεδρίαση θα μας ενημερώσει για το τι συνέβη εκεί. Περάμε στο σημείο 8 αντιπροσωπείς ad hoc στην Οτάβα και στο Μόντρεαλ του Καναδά. Συναντήσεις έγιναν 21 με 23 Μαρτίου του 2016 και εγώ ως πρόεδρος ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής ad hoc. Είχαμε πολύ σημαντικές συναντήσεις και ενδελεχείς συζητήσεις στην ΟΤΑΒΑ με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και πολλοί εκπρόσωποι οργανώσεων κοινωνία των πολιτών εκδήλωσαν επιθυμία συνάντηση μαζί μας. Επίσης συναντήκαμε και με εκπροσώπους γεωργικών συμφερόντων και Ευρωπαίους και Καναδούς και με εκπροσώπους διάφορων καναδέζικων οικονομικών κύκλων. Συζητήσαμε με εκπροσώπους των συνδικάτων του Καναδά. Ε, συναντήσαμε την κυρία Φρίλαντ, την Καναδέζα Υπουργό Εμπορίου και εκεί είχαμε πολύ διεξοδική συζήτηση μαζί της και επίσης συζητήσαμε και με τους ομολόγους μας από την Καναδική Βουλή. Δυστυχώς, την δεύτερη μέρα, 22 Μαρτίου, λάβαμε τα δυσάρεστα μαντάτα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και συγκινήθηκα κι εγώ από το ενδιαφέρον που έδειξαν και την συμπαράσταση και τα συλληπιτήρια των Καναδών. Κρατήσαμε και ένας του και η αρμόδια εμπορίου και πολλοί πολιτικοί από τον Καναδά εξέφρασαν τα βαθύτατα τους συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή τους ε, με σύστιες ε, ε, και μάτιζαν οι σημαίες στον Καναδά, κάτι που δείχνει πόσο συμπάσχει η χώρα αυτή με τα δεινά που έπληξαν την Ευρώπη εξαιτία των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το δεύτερο τμήμα της αντιπροσωπείας έλαβε χώρα στο Μόντρελ. Και εγώ, επειδή είχα μια μικρή εγχείρηση να κάνω Βλέπετε τον επίδεσμο στο χέρι μου. Χρειάστηκε να γυρίσω. Η κυρία Σχάκεν έλαβε τη σκητάλη και ήταν επικεφαλής στο δεύτερο αυτό τμήμα της επίσκεψης. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί ένα μέλος αντιπροσωπείας μας ήρθε μόνο στο Μόντρελ και απουσίαζε από την Οτάβα. Και όσο εμείς ήμασταν στην Οτάβα, ο βουλευτής έδωσε συνέντευξη τύπου, στο μόντραλ, Κάτι που τάραξε τα νερά κάπως στον καναδικό τύπο με αποτέλεσμα μία υπουργός της κυβέρνησης του Κεμπέκ και μία ε, εταιρεία του Καναδά να αρνηθεί συναντήσει μαζί μας εξαιτίας των δηλώσεων που έκανε αυτό το μέλος αντιπροσωπείας που έκανε δηλώσει ε, είτε προσωπικέ είτε εκ μέρους ομάδας που δεν θα έπρεπε όμως σε καμία περίπτωση να δεσμεύουν την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν αρκετά καθόδης η κατάσταση. Πάντως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη συμπεριφορά των Ευρωβουλευτών σε αυτές τις αντιπροσωπείες το διοντολογικό κώδικα που θα πρέπει να ισχύσει σε τέτοιε περιπτώσει. Πιστεύω ότι τα μέλη τη αντιπροσωπεία θα πρέπει να εκφέρουν τι απόψει του ε, ω μέλη τη αντιπροσωπεία και να κρατούν μια συσπηρωμένη συμπεριφορά. Όταν εκφέρουν προσωπικέ γνώμε, να το δηλώνουν και να το ξεκαθαρίζουν. Δεν μπορούν να εκφέρουν προσωπικέ γνώμε δεσμεύοντα το σύνολο τη αντιπροσωπεία. Επίσης, Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δεχθεί αδιαμαρτύρητα τον κατάλογο με ομολόγους ή συνομιλητές, γιατί προσωπούμε διαφορετικές πολιτικές ομάδες και δεν θέλαμε κανένα να μας επιβάλλει τους συνομιλητές μας ή να μας ε, υποδεικνύει ποιους θα συμπεριλαμβάνουμε εμείς στην αντιπροσωπεία μας. Αυτά. Πάντως γενικά ήταν ε, πολύ επικοδομητική και καρποφόρα αυτή η επίσκεψη στον Καναδά. Επί της ουσίας ε, μιλήσαμε κυρίως για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά δηλαδή, που έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 29 Φεβρουαρίου. Έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Διαπιστώσαμε ότι το κείμενο αυτό έχει τροποποιηθεί κυρίως ως προς το θέμα των ανεξάρτητων δικαστηρίων υπάρχει μια θετική εξέλιξη και από καναδικής πλευράς και είναι σπάνιο να έχουμε τόσο θετικά σχόλια, γιατί συνήθως ήταν μορφές αυτές που ακούγαμε. Υπάρχει βέβαια το θέμα της ε, μετα, μεταφοράς των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θέσαμε και μια ερώτηση για τον τομέα των υπηρεσιών. Θα συνεχιστούν αυτά τα θέματα και θα συζητηθούν διεξοδικότερα και με την ευκαιρία της κύρωσης. Πάντως φαίνεται ότι οι περισσότερες πολιτικές ε, ομάδες στον Καναδά είναι υπέρ της ε, συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ της συμφωνίας ΣΕΤΑ δηλαδή. Πάντως έχω την αίσθηση ότι ακολουθούμε παρόμοιες διαδικασίες με τον Καναδά, κάτι που διευκολύνει τα πράγματα. Ακούσαμε βέβαια πολλές επικρίσεις ε, από τους Καναδούς για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πάντως οι Καναδοί έχουν το δικό τους ε, νομικό, δικαστικό και οικονομικό σύστημα που είναι τελείως διαφορετικό από τα Ηνωμένα Πολιτείων και αυτό το επισημάναμε επανειλημμένως. Ευχαριστώ η Τζουντ. Ήθελα να σας πω ότι εκτός από αυτό που είναι την προσωπία θα πρέπει να καταφέρουμε στα πρακτικά ότι όταν κάτι τρομερό γίνει στην ε, πατρίδα μας και στη γενετηρά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κανεί, δεν μπορεί να βρεθεί κοντά στους ε, δικούς του και ακριβώς όλα αυτά τα μηνύματα αλληλεγγύης ήταν πάρα πολύ συγκινητικά αυτά δηλαδή όλα τα, τα, τα μηνύματα αλληλεγγύης από τον Καναδά, από τους εταίρους μας σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και τότε που εμείς ήμασταν στον Καναδά τα πράγματα που ήταν καθόλου ρόδινα οπότε νομίζω ότι αυτό σημάδεψε αυτή την αποστολή και την προσωπία μας επίσης ε, είχε και πολιτικό χαρακτήρα και όχι μόνο χαρακτήρα εμπορική πολιτικής γιατί πρόκειται για αυτές τις ε, αξίες για την ανοιχτή κοινωνία μας την ανοιχτή οικονομία και ακριβώς ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά προβλήθηκαν εντυπωσιακά και επίσης είχαμε και κάποιες επικρίσεις ε, κατά την αποστολή και πρόκειται για κάποιες επικρίσεις για την των πολιτών ε, στην Ευρώπη σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες για τη νέα, νέα γενιά. Συναντήσαμε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και μας είπαν τις ανησυχίες τους Οπότε θα πρέπει φυσικά όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη όταν ήρθε η ώρα συζήτηση για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ του αμέσω επόμενου μήνε. Μια που δεν ήρθατε στο Μόντρελ, ήμουν εγώ και νομίζω η μόνη που παρίσταται από τους βουλευτέ παρέστε στο Μόντρελ και παρά όλε αυτέ τι εντυπωσιακέ δημοσιεύσει στον τύπο ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικές παραγωγικές συνεδριάσεις με τις ε, αρχές ε, του Μοντρέλ του Κεμπέκ, με τοπικούς άρχοντες και οπότε δεν μπορούσαν να μας εκτρέψουν του σκοπού μας όπως κάποιοι προσπάθησαν και νομίζω ότι περισσότερο σαν άτομα παρά σαν ομάδα προσπάθησαν πάρα πολύ και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε, να προβληματίσει και θα πρέπει να συζητηθεί αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο για το τι θα γίνει με τις μέλουσες αντιπροσωπείες. Πάντως, νομίζω ότι η συμπεριφορά κάποιου συγκεκριμένου συναδέλφου ε, δεν δυναμίτησε το συμφέρον του Κοινοβουλίου. Στο Μόντριο τέλος πάντων ήταν η υποδοχή μας πάρα πολύ θετική, ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις ε, με τους επισήμους εκεί στο Κεμπέκ. Αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να σου το πω, μια που παρέστην εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλά λοιπόν, το υπαριθμόν 9. Η ειδική αντιπροσωπεία για τον Ισημερινό. Εκ με την αντιπροσωπεία στον, Καναδό, στον Καναδά, συγγνώμη, ε, μετέβηκε αντιπροσωπεία στον Ισημερινό, στο Εκουαδόρ για να συζητήσει θέματα εντάξει στις χώρες αυτής στη Συμφωνία Κολομβίας-Περού με μέλη τους κυρίους Φίσας και Σόλτς. Ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σόλτς, αλλά είναι απόνα. Κύριε Φίσας, αρχίστε εσείς τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θα μιλήσει ο κύριος Σόλτς. Ε, αλλά καλύτερα από μιλόγω για να φύγω. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή η αποστολή στο Εκουαδόρ. Ε, υποφαινόμως ο κύριος ε, ε και άλλοι. Και έχω να σας πω τα εξής. εγώ δεν ξέρω, έχω να πω ότι έχουμε μια συμφωνία γέννη και συστήμα γεννημένων προσθέσεων συν και είχαμε τη συμφωνία η οποία έλεγε ε, το 14 τον Οκτώβριο και ε, μετά ανανεώθηκε η συμφωνία αυτή για δύο χρόνια. Λίγη φέτος όπως προέβλεπε και δέχεται το Εκουαδόρ για αυτή τη συμφωνία του ελεύθερου εμπόριου, είναι να γίνει μια συμφωνία σαν και αυτή που ισχύει για Κολομβία και Περού. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία ε, είχαμε δύσκολες διαπραγματεύσει, αλλά είπαμε ότι στον σημερινό θα πρέπει όπως οι, οι, οι γειτονικέ χώρε να δεχθούν την προσχώρηση του σημερινού εις αυτήν την Συμφωνία Ελευθερών Εμπορίου. Πάντως προκλήθηκε κάποια καθυστέρηση, δεν ξέρω τώρα, ε, ίσως ήταν λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά πάντως τελικά υπήρξε έγκριση από πλευρά τη Επιτροπής και κατόπιν το Συμβούλιο όπως συνήθως είπε για προθεσμία εξαμήνου, ούτως ώστε να γίνει η οριστική έγκριση. Και κατόπιν θα πέρασε συμφωνία από το Κοινοβούλιο. Και ίσως επομένως έτσι 31 Δεκάτου του 16 να μην έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι η τελευταία μας ε, ολομέλεια θα είναι στις 12 ε, Δεκεμβρίου. Αυτό δεν θα διευκολύνει τα πράγματα για τον εσημερινό. Γιατί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρώσουν ε, τους σχετικούς δασμούς. Οπότε οι αρχές της χώρας ξέφρασαν τις ανησυχίες τους, συζητήσαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πολλούς υπουργούς. Αλλά και με των πολιτών, με επιχειρηματίες, με κάποιους ε, φορείς του ε, θα πληθυσμού και είπαμε ότι πέραν των δισταγμών θα πρέπει να συναυθούν αυτές οι σημαντικές ε, συμφωνίες που είναι τόσο σημαντικές για τη χώρα και ως ε, Κορέα βέβαια κατέβησε κατέβει σε εκλογές ε, αρχές του 17 οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτή η συμφωνία ελευθερών εμπόριο. Οπότε μας είπαν ότι ανησυχούν πάρα πολλοί οι συνομιλητές μας φοβούνται πως δεν υπάρχει μέχρι τέλος του έτους έγκριση, αλλά είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε την περνάει από το χέρι μας, ούτω ώστε να συντιμήσει τις σχετικές προθεσμίες του Συμβουλίου, που εξάμεινο να γίνει ας πούμε τρίμηνο, ούτω ώστε να τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί και έτσι να γίνει η έγκριση από το Κοινοβούλιο πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2016 ο τύπο τη κυβέρνηση του σημερινού είπε ότι προτίθεται να έρθει εδώ να συναντήσει ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και ο κύριος Σόλτ κάλεσε τον Υπουργό Διεθνού Συμπορίου να έρθει στην Επιτροπή μας τον Απρίλιο, στην συνάντησή μας. Οπότε θα έρθει και θα μας διατυπώσει τις ανησυχίες του. Σύμφωνα με απόλυτα με τον κύριο Σόλτ, να πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, το ώστε τα πράγματα να διευκολυνθούν και να έχει υπογραφεί συμφωνία πριν την 31η Δεκεμβρίου. Θα πρέπει επομένω να έρθουμε σε επαφή με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιμείνουμε οι προθεσμίες να γίνουν συντομότερες. Δεν υπάρχει κάτι να ζητηθεί. Η ουσία του θέματο έχει κλείσει, έχει συμφωνηθεί. Όπω ξέρετε είναι πολύ περίπλοκη η οικονομική συγκυρία στη χώρα. Έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει πρόβλημα και με τις εξαγωγές και υπάρχουν κάποιοι δασμολογικοί φραγμοί όσον αφορά κάποια ευρωπαϊκά προϊόντα. Εμεί, αυτό το καταγγείλαμε. Και ένα συγκεκριμένο δασμό ε, που αποσκοπεί στο να εμποδίσει αγωγέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι κατά των όσων ε, προβλέπει ο ΠΟΕ. Αυτό είναι παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να δείχνουμε κάτι το οποίο είναι κατά του ΠΟΕ. Το με αυτό προς τις ε, αρχές της χώρας. Και το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ένα plan B ε, και να έχουμε κάποιο είδους παράταση της ισχύω της συμφωνίας. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα διευκολυνθούν οι πραγματεύσεις και θα κλείσει συμφωνία μέχρι τα τελή του έτους πρόεδρος. Δεν ε, νομίζω να υπάρχει καμιά αντίρρηση σε αυτό που είπατε, δηλαδή να περαιτέρω δραστηριοποίηση. Χέλμουτ, εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Θα είμαι σύντομο και θα συμπληρώσω μόνο τα δηλαδή, ορισμένα στα όσα είπε ο συνάδελφός μου Φίσας. Αναφέρθηκε σύντομα στην δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, του σημερινού δηλαδή, ε, οικονομία που εξαρτάται από το δολάριο και καθώς πέφτει και η τιμή του πετρελαίου αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές και ενδογενείς προκλήσεις διότι άλλωστε υποτιμήθηκε και το κολομβιανό νόμισμα κατά 60%. Η εξισορρόπηση μέσα από το φάσμα των εξαγωγικών προϊόντων αναγκάζει τώρα τον Ισημερινό να γίνει ιδιαίτερα επινοητικός για να μπορέσει να υπερβεί τις δυσκολίες αυτές, ιδίως και απέναντι στην πρόκληση τι θα συμβεί μετά τη λήξη, μετά δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου του 2016, όταν θα επιβληθούν δηλαδή οι δασμοί στα εξαγώγημα προϊόντα που εξαγόνται στην Ένωση. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση όλοι οι συνομιλητές μας από τις μεγάλες ενώσεις οικονομικών φορέων μέχρι τις μικρές ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις τομεακές οργανώσεις των όσων απασχολούνται στην βιώσιμη μικρή οικονομία από παραγωγούς δηλαδή ε, καφέ μέχρι μπανανών Όλοι μας εξήγησαν ότι η ίδια ύπαρξη των επιχειρήσεών τους διακυβεύεται. Έχουμε λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα μπροστά μας και πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανάγκες αυτές του σημερινού για να ασκήσουμε και πίεση στο Συμβούλιο Υπουργών. Μπέντ, εσύ ως πρόεδρος και εμείς ως εισηγητές μπορούμε να συντάξουμε επιστολή προς την Ολλανδική Προεδρία και να την παρακαλέσουμε Εν ώψη του ιστορικού αυτού των ε, εξελίξεων δηλαδή, της πραγματικής οικονομίας στον Ισημερινό να λάβει τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε να ασκήσουμε και εμείς τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και να μπορέσουμε να ε, ελέγξουμε την συμφωνία ήδη πριν από το τέλος του έτους. έτσι ώστε η συμφωνία να στηρίξει την πορεία του σημερινού προς μια βιώσιμη οικονομία. Έχουν ήδη σημειώσει επιτυχίες, άλλωστε και στην Επιτροπή Σχεδιασμού της, της κυβερνήσεως του Ισημερινού, εκεί δηλαδή είχαμε προσκληθεί και μπορέσαμε να συζητήσουμε μαζί τους έκαναν, έχουν ακολουθούν και αυτή την πρακτική των μελετών αντικτύπου για να δουν ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στους επιμέρους τομείς της οικονομίας τους. Τονίζω επίσης ότι βέβαια μιλήσαμε πράγματι με πολλούς υπουργούς αλλά και στην Βουλή του Ισημερινού συναντηθήκαμε με την αναπληρώτρια πρόεδρο της Βουλής τους και με αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων της η σημερινή έθνοσυνέλευση, και μας δήλωσαν και αυτοί ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, από τις κοινοβουλευτικέ τους ομάδες, ώστε το αργότερο, τον Οκτώβριο τρέχοντος, να μπορέσει να γίνει κύρωση της συμφωνίας από την Βουλή του Ισημερινού. Να υπάρξει δυνατότητα δηλαδή να τοποθετηθούμε ταυτόχρονα επί της ε, συμφωνίας. Ταυτόχρονα δεχθήκαμε την πρόκληση, ενδεχομένως δέχθηκαν αυτή την πρόκληση, να έρθουν εδώ, να ε, μας επισκεφτούν με τον Υπουργό. Άρα δηλαδή εκπρόσωποι και της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας της χώρας και σε αναλογία, κατά αναλογία συζητήσαμε και με πάρα πολλές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μαζί και με, με ποικίλου εκπροσώπους του ηθαγενούς πληθυσμού οι οποίοι μας εξήγησαν ποιες είναι οι επιφυλάξεις τους ότι φοβούνται δηλαδή ότι αυτοί η βιώσιμη ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ενδέχεται να υποστεί βλάβη από την διμερή συμφωνία. Ιδίω δε ο αγροτικό τομέα, τα προϊόντα του αγροτικού τομέα, καθώ και η εξορρυκτική βιομηχανία που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την βάση της απασχόλησης του Ιθαγενούς πληθυσμού και ότι αυτά μπορεί λοιπόν να τους στηρίξουν πολλέ δυνατότητε. Δεν θεωρούν λοιπόν πολιτικά ότι μπορούν να στηρίξουν τη συμφωνία αυτή. Προσπαθήσαμε να συναντηθούμε λοιπόν με εκπροσώπου όλου του φάσματος. Θα υποβάλουμε πλήρη έκθεση, άλλωστε είμαστε στη διάθεσή σα για να σας απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Δεν θέλω να παραλείψω δε, εν προκειμένου, να ευχαριστήσω και τον πρέσβη Πέτερ Σφάιγερ, και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για την πραγματικά εξαιρέτη στήριξή τους, καθώς επίσης και τις δύο διερμηνείς μας, κυρία Πίτερσεν και κυρία Ιμπαρό, οι οποίες εργάστηκαν δίπλα μας επί 18 ώρο. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής, ιδίως τον Μάρκ, για την θαυμάσια προετοιμασία αλλά και υποστήριξη προσέφερε στο ταξίδι μας. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλμουντ. Αυτό το τελευταίο το προσυπογράφω ευχαρίστως. Όλα τα ταξίδια αντιπροσωπιών της Επιτροπής μας απολαμβάνουν τον τελευταίο καιρό πραγματικά μια άψογη διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν ε, αγαπητά μέλη της Γραμματείας. Ό,τι αφορά την επιστολή, σύμφωνοι. Να γράψουμε μια επιστολή προς την Ολλανδική Προεδρία και να τη ζητήσουμε να επιταχύνει. Να επιταχύνει, να προλάβουμε τις προθεσμίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά ε, δυσχερής κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο σημερινός. Τώρα, ας ακολουθήσει το θέμα υπαρχών 11 της ημερήσιας διαταξή μας. Α, με συγχωρείτε, ναι. Για το 10 αποστολή στην Τουρκία που προβλεπόταν για 19 έως 31 Μαρτίου ε, για λόγους ασφαλείας ακυρώθηκε. Έχετε βέβαια πληροφορηθεί κι εσείς ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη είναι ιδιαίτερα ανισχυτική μετά από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν εκεί. Ακολουθεί το θέμα υπαριθμών 11. Είχα δει τον αρμόδιο συνάδελφό μου. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Κοιτάξτε. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στην ημερησία διάταξη. Έχουμε ένα πλήθος ε, συμφωνιών που έχουμε συζητήσει ήδη εξωτικά και αν στρέψουμε τα βλέμματα προς τα πίσω από την 1η ε, Δεκεμβρίου του 2009 που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία της Λισαβόνας έχουμε εμείς αρμοδιότητα για ε, επενδυτικές συμφωνίες. Να παρακολουθούμε δηλαδή την εξέλιξη των συμφωνιών αυτών και να τις εγκρίνουμε ή να τις απορρίπτουμε. Το 2012 ήδη εγκρίναμε δύο σημαντικά νομοθετήματα. Αφενός για το λεγόμενο grandfathering των υφιστάμενων διμερών επενδυτικών συμφωνιών με ξεκάθαρη εντολή και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις διμερείς αυτές συμφωνίες όπου στο ενδεικτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδα ότι σκέπτονται για το 2020 να λήγουν αυτές οι συμφωνίες. Μήπως εδώ μπορούν να επιταχύνουν λίγο αυτό, σκέπτομαι εγώ. Και το δεύτερο νομοθέτημα είχε ως εξή εάν γίνει προσφυγή κατά της Ένωσης ή των χωρών μελών, ποιος καλείται να πληρώσει. Ποιο φέρει δηλαδή την οικονομική ευθύνη. Δύο νομοθετήματα, όπως είπα, τα οποία εγκρίναμε το 2012 και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο όπου κανονικά θα πρέπει να μιλήσουμε για το μέσον της επενδυτικής προστασίας και μάλιστα να συζητήσουμε κάπως διεξοδικότερα. Επ' αυτού έχω τώρα πέντε θέματα τα οποία με απασχολούν κάπως ιδιαίτερα. Αφενός, το νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του. Εδώ συναρτάται και η εμπειρία την οποία διαθέτουμε από την επενδυτική πολιτική που ασκήθηκε μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνος. Πού πήγε κάποια, πού πήγαν κάποια πράγματα καλά, πού πήγαν λιγότερο καλά, ποιες είναι οι προκλήσεις. Και τρίτο, να δούμε τι γίνεται και με τον χάρτη ενέργειας. Θα θυμάστε ότι ο χάρτης ενέργειας είναι και η μοναδική σύμβαση που σύναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, με το ISTS. Εδώ δεν ευθυνόμαστε εμείς. Αυτά νομίζω έχουν γίνει ήδη από το 1994, όταν δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν είχε ακόμα σχετική εξουσία, όπου ήταν όμως η πρώτη και μοναδική συμφωνία που διέθετε ISTS, δηλαδή Σύστημα Επίλυσης Διαφορών Επενδυτού Κράτους. Ως τώρα υπάρχουν 89 υποθέσεις ωστόσο που βασίζονται στον χάρτη ενέργειας. Άρα είναι σκόπιμο να αναλογιστούμε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, ιδίως διότι στο μεταξύ έχει προχωρήσει η συζήτηση από το 1994 βέβαια, και η πρόταση για ένα σύστημα ICS κινείται προς άλλη κατεύθυνση και το ερώτημα είναι δεν θα πρέπει στον χάρτη ενέργειας να ενσωματωθεί και το σύστημα ICS. Τέταρτο, τι γίνεται με τις ε, συμφωνίες, με τις διμερείς ε, επενδυτικές συμφωνίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταξύ χωρών μελών. Ε, υπάρχουν εκεί διατάξεις ISTS. Το δε πέμπτο θέμα που με απασχολεί, τι γίνεται με τις συμφωνίες χωρών μελών έναντι τρίτων χωρών. Μήπως πρέπει να ζητήσει δεσμευτικά συστήματα ACS η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτού του grandfathering. Α, πέντε ερωτήσεις λοιπόν που με απασχολούν και ελπίζω να ακούσω κάποιες απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, να δώσω κάποιες αρχές απαντήσεων έσω στα θέματά σας. Κάτω των όσων μας είπατε για αυτήν την ανακοίνωση για την εμπορική πολιτική, αλλά και το πρόγραμμα εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς έχει τοποθετηθεί ότι θα, θα έπρεπε κατά αυτή τη θητεία να εξετάσουμε ξανά την εμπορική πολιτική. Και ε, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η προβληματική τώρα. Γιατί πολλά από τα θέματα τα οποία θίξατε ε, βεβαίως ε, και εμά μας απασχολούν. Οπότε πρώτα πρώτα να σας πω δύο λόγια για το νομικό πλαίσιο. Όντω έχουμε αυτού τους δύο βασικούς κανονισμού και να σας πω δύο λόγια για το πώς λειτουργούν. Κάτι το οποίο ήταν το δεύτερο σημείο το οποίο εσεί αναφέρατε. Πάντως η γενικότερη εντύπωση που έχουμε είναι ότι γενικώ αυτή η μεταβατική περίοδος ήταν αρκετά ομαλή και υπάρχει και ένα νομικό σημείο το οποίο μα απασχόλησε και όχι τόσο ω προ το Συμβούλιο αλλά ως προς τα κράτη-μέλη. Ακριβώς ε, αυτό καλύπτει το άρθρο 207. Αυτό το ζήτημα του FDI, δηλαδή του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε αυτό και θέλουμε να επανέλθουμε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι το άρθρο του 207 ομιλεί περί εξωτερικών ε, επενδυτών, αλλοδαπών επενδυτών. Και βέβαια ε, για την περίπτωση της Σιγκαπούρης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από εδώ υπάρχει και αρμοδιότητα ε, γιατί έχει σχέση και με τα άρθρα 63 66 για την κίνηση κεφαλαίων. Ό,τι καλύπτεται δηλαδή από αυτά τα άρθρα ε, ό,τι ισχύει ιστορικά και εξωτερικά, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του TFU. Πάντως, αυτά τα μέτρα, από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, έχουν αποδώσει. Και έχω να σας αναφέρω παραδείγματα. Πρέπει να συζητηθούν και οι συνέπειες αυτών. Τότε πώς να ισχύει αυτός ο κανονισμός για το Grand Father και μέχρι το 2015 είχαμε 80 εγκρίσεις αδειοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει τον λογοκανονισμό και οπότε ε, εγκρίθηκαν κάποιες ε, διαπραγματεύσει και είχαμε 36 αποφάσεις που δώσαμε πράσινο φως και επίσης δώσαμε πράσινο φως και για νέες διαπραγματεύσει πολλές από αυτές τις αποφάσεις αφορούσαν και κάποιες συμφωνίε των οποίων διαπραγματεύσει εκκρεμούσαν πριν την αναξίσκευση του οργανισμού. Και όπως σας είπα έχουμε συνολικά 80 θετικέ ε, αποφάσεις. αλλά είχαμε και άλλες οι οποίε εκκρεμούν, δεν έχουν ακόμα κρυθεί. Και είπαμε σε σχέση με αυτά ότι τώρα έχουμε ε, το θέμα της μεταρρύθμισης και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις συζητήσεις και γι' αυτό και δεν αποφασίσαμε τίποτα. Ε, έρθουμε πρώτα να ξεκαθαριστεί πώς θα δημορφωθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογα θα ενεργήσουμε για αυτές τις εγκρίσεις. Εκεί που δεν δώσαμε έγκριση ε, ήταν διότι υπήρχε αντίθεση ως προς τον κανονισμό. Δηλαδή δεν συνάδουν αυτές οι περιπτώσεις με την πολιτική μας ή τέλος πάντων ήταν ε, ε, αντίθετες προς κάποιες ληφθήσεις ήδη αποφάσεις. Υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Παρ' όλα αυτά, είναι ψηλό ο αριθμό των εγκρίσεων, αλλά 40% των εγκρίσεων που δώσαμε δεν αφορά νέες συνθήκες, ε, αφορά κάποια πρωτόκολλα ε, τροποποιητικού χαρακτήρα ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν υπάρχουσε συνθήκες με τη σχετική νομολογία. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με ε, τις ε, εξαιρέσεις προς ήδη σχείοντες κανόνες. Υπήρχε ένα κενό μετά την ε, θέση της ε, συνθήκη της Λισαβόνα. Προσπαθήσαμε να δούμε τι θα κάνουμε και άρχισε μια ματιά στο τι γίνεται με τις παρούσες διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε τις περισσότερες κρίσεις. Τι γίνεται με τις διάφορες συμφωνίες, με συμφωνίες ελευθερών εμπορίου και οπότε έχουμε 200 ε, τροποποιήσεις συμφωνιών εμπορικών. Οπότε δεν μπορεί να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να εκτελεστούν οι διαμοντευτικέ εντολές ακόμα και σε διμερές επίπεδα. Τότε θα υπάρχει περισσότερη εναρμόνιση, περισσότερη συνέπεια μακρόπνοη. Ακόμα επομένω δεν ολοκληρώθηκε η προσπάθειά μας, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και όλε οι νέε συμφωνίε που έχουμε διαπραγματευτεί και που πρόκειται να κυρωθούν θα αφορούν ακριβώς την αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνίων γιατί έχουμε πάρα πολλές α, διμερείς συνθήκες των κρατών μελών που θα πρέπει να φροντίσουμε για να συνάδουν με την πολιτική μας. Κάτι άλλο το οποίο θίξατε πρόεδρε είναι για τη συνθήκη που αφορά τον ενεργειακό χάρτη. Αυτό έχει σχέση και με τις διμερείς συνθήκες της εσωτερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε να δούμε τι εμπειρία έχουμε αποκτήσει, τι γίνεται από τα κράτη-μέλη, αλλά πρώτα-πρώτα θα πρέπει να σας αναφέρω ότι η σχετική συνθήκη όπως και εσείς αναφέρατε ε, ανάγεται στο 1994 και τότε όλοι θεώσουν ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σύγχρονο ο σκοπός τότε ήταν να έχουμε μια σφαιρική προστασία. Και από τη μια μεριά είχαμε την ασφάλεια δικαίου στην Ευρώπη, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, και από την άλλη μεριά είχαμε την CIS. Και είπαμε ότι από την άλλη μεριά θα έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά ε, για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές από τη από το μετασχηματισμό στην Ανατολική Ευρώπη, σε εκείνες τις χώρες. Τώρα κάπως τα πράγματα άλλαξαν και είχαμε πάρα πολλές υποθέσεις, είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτός ε, της, ε, του αρχικού μας σκοπού, αλλά εμπίπτουν στους βασικούς κανόνες προστασίας στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη η συμφωνία είναι για πέταμα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε η χρησιμότητα της συνθήκης εκείνης. Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα τώρα και νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει. Ποιο είναι το θέμα αυτό. Τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση. Και το τοπίο πώς έχει διαμορφωθεί, πώς έχει εξελιχθεί σε σχέση με τον χάρτη των ενεργειακών. Βεβαίως και αυτό μας απασχολεί. Και άλλοι ασχολούνται πάντως με το ίδιο θέμα. Θα πρέπει όμως και εμείς να αντιμετωπίσουμε το τι θα γίνει. Και συζητήσαμε με την γραμματεία του Ενδιακού Χάρτη. Σήμερα πάντως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ήδη είπαμε ότι έχουν αλλάξει κάποιοι ορισμοί και είπαμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η συνθήκη του Ενδιακού Χάρτη, να έχουμε πολυμερή προσέγγιση σε σχέση με τη νέα πολιτική μας. Πρόκειται όμως για μακρόπνο στόχο και θα πρέπει να μας βοηθήσουν και άλλοι σε αυτή μας την προσπάθεια. Γιατί ακριβώς στην γραμματεία έχουμε ε, χώρες με τις οποίες έχουμε κάνει παρελθόν διαπραγματεύσεις χώρες όπως η Ιαπωνία. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις χώρες. Άρα διερευνούμε το τι δυνατότητες υπάρχουν. Είναι σαφής η στόχη μας. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω τίποτα, ακόμα τα σκεφτόμαστε. Και όπως γνωρίζετε, ακόμα δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής. Υπάρχει πάντως η εντολή για να θεωρηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως κάτι γίνεται, δεν βρισκόμαστε στο α, στο 0. Να δούμε και πώς θα συνοηθούμε και με την ε, ε, Ιαπωνική Προεδρία ε, της Γραμματείας του Φορέα της ενεργή, του Ενεργείου Χάρτη. Και το επόμενο κύριε Πρόεδρε, το οποίο θέλατε να συζητήσουμε Θέλατε να δούμε τι γίνεται με τις διμερείς εμπορικές συνθήκες στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξέρετε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα και ότι δεν θεωρούμε ότι αυτές οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να συνυπάρχουν με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε αρχίσει ε, να κινούμε την διαδικασία επί για πέντε τουλάχιστον κράτη-μέλη. Και μιλούμε για περίπου 200 ε, τέτοιες επενδυτικές συμφωνίες ε, και ε, σταθήκαμε σε μια-δυο από αυτές να δούμε τι θα κάνουμε. Τα δε κράτη-μέλη έχουν ε, μια ποικιλία τοποθετήσεων αλλά βέβαια κατάσταση μέχρι ένα σημείο είναι δύσκολη αλλά κάποια κρατημέλη επίσης ε, σαφώς βλέπουν ότι θα πρέπει κάπως να βοηθήσουν και να δοθεί κάποια συνέχεια στην πολιτική. Έχουμε και επίσης και τους ανθρώπους της Αρμόνας Γενικής Διεθνής με τους οποίους προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα πρόβλημα, διότι με τις επαφές μας με το Συμβούλιο δεν έχει ξεκαθαριστεί από νομική πλευρά τι είναι δυνατόν να γίνει. Υπάρχει πάντω αυτή η επικάλυψη με κάποιε διατάξει τη συνθήκη. Εκεί οι επαφέ, στο Συμβούλιο δηλαδή, έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Δηλαδή λέμε, αν δεν υπάρχει σχετική προστασία, τη ρύθμιση, τι θα κάνουμε, γιατί σε πολλέ περιπτώσει. να υπάρχει νομική κάλυψη είναι χρήσιμο ή τώρα θα πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε αφού δεν έχουμε ένα πλήρε σύστημα επενδυτικών διμερών συμφωνιών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί για του επενδυτέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω κάποια κρατημέλη θα αναζητήσουν εναλλακτικά μέσα και εναλλακτικέ διαδικασίε. Σύντομα πιστεύω ότι κάτι θα βγει από αυτή την προσπάθεια. Και τώρα, το τελευταίο σας ε, θέμα που επίσης είναι πολύ σημαντικό, ποια είναι αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης. Τι γίνεται με τις συμφωνίες, τις επενδυτικές με τρίτες χώρες. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές από αυτές τις αναδιαπραγματεύσεις ξεκίνησαν από το ότι ζητήσαν τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τις σχετικές συνθήκες. Σας είπα για την περίπτωση της Νομισματικής Ένωσης. Εκεί που είχαμε κάποιες παραβιάσεις στις ε, σχετικές ρυθμίσεις. Γιατί εκεί είχαμε κάποιες ρήτρε που προέβλεπαν για κινήσεις κεφαλαίου και σε περιπτώσεις εκτός εκτάκτων γεγονότων. Οπότε είπαμε τώρα ότι θα πρέπει να γίνουν διάφορες αλλαγές να δούμε τι θα γίνει ας πούμε με τις κρατικές ενισχύσεις από το TTIP θα δείτε το πώς δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιες ενισχύσεις αλλά έχουμε και άλλα θέματα τα οποία είναι πιο, πολι... πιο πολιτικού χαρακτήρα δηλαδή τι εγκρίσεις θα πρέπει να στο μέλλον ακόμα και δεν είναι κατά της ε, νομής τάξης, αλλά είναι κάτι που αντιβαίνει στην ε, επενδυτική πολιτική. Ας πούμε υπάρχει κάποια συμφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με το TTIP και για τις άλλες διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για να έχουμε ε, ένα σύστημα που θα αντικαταστήσει για τις επενδύσεις την διατησία. Για αυτές τις ε, συμφωνίες, σε αυτές δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε μέχρι πού θα προχωρήσουμε και άρα αυτό και μελετούμε. Τι θα προβλέπει η πολιτική που τώρα χαράσεται. Ξέρω ότι δεν συμφωνείτε όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά τουλάχιστον κάποιες περιοχές του Κοινοβούλιο συμφωνούν με την ε, πολιτική μας, την οποία και τώρα μελετούμε. Και στο μέλλον πάντως θα δούμε τι θα γίνει, με συγκρίσεις που να δώσουμε. Ακόμα δεν έχω τίποτα οριστικό να σας αναφέρω. Α, εδώ θα βάλω όμως τελεία. Βεβαίως και μπορούμε να συζητήσουμε κι άλλο. Αλλά να μην με Περιμένω να ακούσω τη γνώμη σας και ό,τι ερωτήσει έχετε θα προσπαθήσω να τι απαντήσω. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Οι σοσιαλιστές πρώτοι, Τζουτ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Ένα γενικό σχόλιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα επενδυτικής πολιτικής, στη συζήτηση για την επενδυτική πολιτική. Μετά τις ε, ε, ανησυχίες που εκδηλώσαμε και εμείς και στη, συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση που έγινε για τις επενδυτικές συμφωνίες και συνθήκες. Αυτό δείχνει ότι όταν κανείς ε, επισημαίνει ανησυχίες ε, και αυτό γίνεται σε ευρία κλίμακα, παρακινεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι μεταρρυθμίσεις. Και στα πλαίσια τη πρόοδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, καλό είναι να το θυμόμαστε. Μερικέ φορέ χρειάζονται πολιτικέ κρίσει για να μεταρρυθμιστούν πολιτικέ. Αυτά ω γενικό αρχικό σχόλιο. Βέβαια, ακόμη έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε σε ό,τι αφορά την επενδυτική μα πολιτική. Και έχω δύο ερωτήσει. Ερώτηση πρώτη. Η ρήτρα των κεκτημένων δικαιωμάτων, grandfathering ε, και η σχετική νομοθεσία λέει ότι όταν μια Ευρωπαϊκή Επενδυτική Συμφωνία αντικαθιστά ε, διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Στις περιπτώσεις που εξετάζεται τώρα, ε, επενδυτικές συμφωνίες που περιμένουν κύρωση, έχει μια επισκόπηση πόσες φορές ε, αντικαθιστούνται ε, Τέτοιε ε, επιλύσεις διαφορών μεταξύ των κρατών από επιλύσεις διαφορών κράτου επενδυτή. Γιατί σε πολλέ διμερεί επενδυτικέ συμφωνίε έχουμε συστήματα επιλύση διαφορών μεταξύ κρατών. Κυρίω οι παλιότερε επενδυτικέ συνθήκε. Οι νεότερε συνθήκε έχουν ISDS, δηλαδή επίλυση διαφορών κράτου επενδυτή. Αυτό που με ενδιαφέρει. Γίνεται μια αναβάθμιση, γίνεται αλλαγή και αντικατάσταση του ενό από το άλλο μέσω των ευρωπαϊκών επενδυτικών συνθήκων και συμφωνιών. Σε ό,τι αφορά τις επιλύσεις διαφορών ε, μεταξύ κρατών, κράτους-κράτους, πολύ δώρος γίνεται για την επενδυτική πολιτική και κυρίως για τα προβλήματα που δημιουργεί η επίλυση διαφορών κράτους-επενδυτή. Αυτό έχουν επισημάνει ε, δικηγόροι που ασχολούνται κυρίως με τις επενδύσεις, που μιλούν για το ρόλο του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου που θα πρέπει να αναβαθμιστεί καθώς και του συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ των κρατών. Η Γενική Διεύθυνση Trade ε, το έχει αυτό το θέμα καθόλου στη, στο πρόγραμμά της ή θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό αντί να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό διεθνές δικαστήριο, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους υπάρχοντες ε, νομικούς μηχανισμούς για να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε στην ευρωπαϊκή επενδυτική πολιτική. Ευχαριστώ. Κανένας από το, από το ECR, την Άλντε, όχι, η Γκουέ, ο κύριο Σόλτς. Και εγώ θα ήθελα να ζητήσω την ενημέρωση. Η Τζουντ ρώτησε, ξέρετε ότι η ομάδα μας θεωρεί προβληματική, ε, προβληματικό το μηχανισμό ISTS και, τον, και τη νέα πρόταση, διότι δεν έχει αλλάξει λογική στην οποία βασίζεται. Και γι' αυτό η ερώτηση, δεν θα πρέπει να επανέλθουμε στο ερώτημα ότι όπως κράτος προς κράτος ή ιδιώτης προς κράτος, αυτό που μπορεί να συζητηθεί, να πάνε στα συνηθισμένα δικαστήρια. Να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η τακτική αυτο που θα να προσφύγουν στη τακτική δικαιοσύνη όπου υπάρχουν διαφορές. Γιατί πρέπει να επινοήσουμε ειδικού κανονισμούς που χορηγούν στους επενδυτές ιδιαίτερα δικαιώματα. Δεύτερο, αυτή η συμφωνία grandfathering, πατρογονικής ρήτρας ή κεκτημένου δικαιωμάτων. Είπατε κι εσείς ότι δεν είμαστε εμείς οι ένοχοι κύριε Πρόεδρε διότι έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. Όμως όταν είχαμε την τελευταία φορά συζητήσει την ε, συμφωνία grandfathering στην προηγούμενη θητεία συζητήσαμε και το θέμα αυτό. Ήδη τότε εδίδεται η δυνατότητα επανεξέτασης αυτής της grandfathering και στα πλαίσια αυτής να θέσουμε στην στόχευση αυτό το σύστημα ISTS, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μια άλλη θέση απέναντι στα συστήματα ISDS και ICS. Τώρα, για την Κίνα. Έρχονται τώρα άλλοι εταίροι με τον παλαιό μηχανισμό, τον οποίο πήραν από εμάς ή από άλλες χώρες του ΟΣΑ και που έχουν συνηθίσει να τον χρησιμοποιούν. Και τι κάνουμε τώρα, πώς τους αντιμετωπίζουμε εμείς αυτού, αυτούς την ώρα που τα αναθεωρούμε. Ενδιαφέρουσα ερώτηση η Γερμανία, για παράδειγμα, ενέκρινε το 2005 συμφωνία με την Κίνα που περιλαμβάνει σύστημα ISTS. Η πράσινη τώρα, η Φραντσίσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Εάν ε, προβληματίζεστε τώρα και με τις χώρες μέλη, να το κάνετε και ευρύτερα. Και ποιες είναι οι αντιδράσεις τους απέναντι στον προβληματισμό σας σχετικά με το ISTS ή άλλες ICS συγγνώμη, ε, και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Για το grandfathering εμείς στείλαμε καταληκτική ρήτρα sunset clause για όλες τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Ποια είναι όμως τώρα η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα που εξακολουθούμε να έχουμε όλες αυτές τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες εν ζωή. Μήπως θεωρείτε ότι ή το λάθος να μην ζητήσετε ε, ρήτρα λήξης για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και πώς αντιδρούν οι χώρες μέλη στις συστάσεις που τους δίνεται για την έγκριση νέων διμερών επενδυτικών συμφωνιών. Τέλος, μια και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την συμφωνία ΣΕΤΑ και την προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν σχετικά με το εάν το ISTS είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης ή μήπως είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα. Η Ίνμα. αρμοδιοτητα ευχαριστω Πρόεδρε. Έχω δύο σχόλια, αφού σας ευχαριστήσω προηγουμένως για την παρουσίαση και την ενημέρωση. Μόλις επέστρεψα από τη Σιγκαπούρη. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ε, ανησυχεί τα μάλα σε σχέση με το άνοιγμα, ε, την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας ε, σε σχέση με την ανάγκη να προσαρμόσουμε το νέο σύστημα στο σύστημα των επενδυτικών δικαστηρίων. Και εμείς είχαμε εξηγήσει την αποστολή αυτή τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπαμε θα ήταν αδιανόητο να στηρίξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία συμφωνία που δεν συμπεριλαμβάνει και το νέο σύστημα. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Η εντύπωση πάντως που αποκόμισα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για το σύστημα και το πώς λειτουργεί το σύστημα και γιατί είναι σημαντικό να το προσαρμόσουμε και να το συμπεριλάβουμε. Ε, εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Δεύτερον, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ της πολυμέρειας. Δεν έχει νόημα η θέσπιση μηχανισμών όπου κάθε ε, συμφωνία διαπραγμάτευσης ε, θα πρέπει να προβλέπει και ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί. Τι στρατηγική θα ακολουθήσετε ώστε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να πρωτοστατήσετε στο σχεδιασμό ενός τέτοιου μοντέλου ομοιόμορφου, ομοιογενούς και δίκαιου για όλες τις χώρες όπου και γίνονται οι επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννη Κλίαρικ. Ε, δεν ε, είχαμε μέλος της ΓΚΟΕ στην αντιπροσωπεία για τον Καναδά, στην αποστολή αυτή ε, είχα την αίσθηση ότι ο Καναδά είναι μια δημοκρατία χωρίς σοβαρό ε, δικαστικό και νομικό σύστημα και ήταν τόσο απαραίτητο να προστατεύσετε τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες απέναντι σε ένα τέτοιο σταθές νομικό σύστημα όπως είναι το καναδικό και γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο να θεσπίσετε ένα νέο νομικό σύστημα ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον πολλαπλασιασμό των επενδυτικών συμφωνιών και συνθήκων, μερικές φορές ε, με σύστημα επίλυση διαφορών κράτου επενδυτή και άλλες φορές χωρί τέτοιο σύστημα, τι γίνεται με την υπόσχεση, την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπέρ ενός πολυμερού συστήματος και για την προστασία των επενδύσεων και των επενδυτών. Γιατί αν έχουμε συμφωνίες αριστερά και δεξιά και δεν είμαστε υπέρ μια συγκέντρωση σε ένα πολυμερές σύστημα, τότε ποτέ δεν θα δημιουργηθεί τέτοιο πολυμερές σύστημα. Επίσης, σήμερα θα πρέπει ήδη να έχουμε κρατήσει μια απόσταση και να μπορούμε να κάνουμε μια πιο νυφάλη αξιολόγηση για το κατά πόσο τα συστήματα με, τις, με επίλυση διαφορών κράτους επενδυτού καθορίζουν τον όγκο των επενδύσεων. Μέχρι στιγμής όλες οι μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι η προστασία των επενδύσεων σίγουρα αυξάνει τον όγκο τους, αλλά καμία μελέτη μέχρι στιγμής, καμία έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει η ύπαρξη ενός συστήματος ISDS προστασίας των επενδύσεων είχε θετικό αποτέλεσμα στον όγκο των επενδύσεων. Και όταν ε, βλέπουμε και τις επενδύσεις στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, χώρα, δεν έχουμε την εντύπωση ότι ο όγκος του σχετίζεται με την ύπαρξη όχι ενός τέτοιου μηχανισμού ISDS. Έχετε εκπονήσει κάποια μελέτη ώστε να γίνεται ένα σχετισμό ή να αποδείξει ότι δεν υπάρχει αντιστοιχεία ή συναφή ε, ε, αιτιότητα σε σχέση με τον όγκο των επενδύσεων και την ύπαρξη ενό συστήματο επίλυση διαφορών κράτου επενδυτή. Έχω και άλλε ερωτήσει, λέει ο πρόεδρο Λάγκε πρώτη συνδέεται με αυτό που έθιξε και ο Γιάννικ. Δεν έχουμε την εντολή μόνο να προστατεύουμε τις επενδύσεις, αλλά και πρόθεση των επενδύσεων. Δηλαδή και να προσέλθουν αλλοδαπές επενδύσεις στην Ευρώπη, αλλά και να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε άλλες χώρες. Διότι αυτό σαφώς ε, συμβάλλει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εδώ ποια είναι η διασύνδεση. Η Υπάρχουν δηλαδή διαρκούς χαρακτήρως ενδείξεις ότι τέτοιοι μηχανισμοί στηρίζουν τις επενδύσεις ή πρέπει να επινοήσουμε άλλες μεθόδους ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια, η επενδυτική προσπάθεια εκατέρωθεν. Εγώ θεωρώ ότι η στάση μας είναι πολύ αμυντική. Δηλαδή προσπαθούμε να επιτύχουμε την υπεράσπιση των επενδύσεων. Όχι τόσο να τις προωθήσουμε με τα αντίστοιχα μέτρα. Δεύτερο, το σύστημα ICS το οποίο συζητούμε είναι όντως ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Βρίσκω εγώ. Ενδέχεται πάντως το σύστημα αυτό να διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο. Εάν συγκρίνω το Βιετνάμ, την συμφωνία ΣΕΤΑ, και την πρόταση TTIP σχετικά με το ICS. Υπάρχουν σε πολλά σημεία ενώ τις τρεις αυτές συμφωνίες σημαντικές διαφορές. Δεν θα τις απαριθμίσω όλες, αλλά υπάρχει ένας αριθμός διαφορών. Έχει κάποιο νόημα όταν δηλαδή έχουμε ως πρόθεση να δημιουργήσουμε ένα διεθνές σύστημα, όπου όμως βλέπουμε ήδη τρεις συμφωνίες που το ρυθμίζουν πολύ διαφορετικά. Εν τέλει, επανέρχομαι στο θέμα της Σιγκαπούρης. Εάν θεωρούσαμε ότι χρειαζόταν κάποια θεμελιώδης αλλαγή στην περίπτωση του Καναδά, τότε κάτι πρέπει να τροποποιηθεί θεμελιωδώς και στην περίπτωση της Σιγκαπούρης. Συζητεί η Κομισιόν με τη Σιγκαπούρη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εσείς κύριε Σλέγεμιλ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και για τις ερωτήσεις. Ε, θα βάλω τα δυνατά μου για να απαντήσω. Θα ξεκινήσω με την συζήτηση της κυρίας Ντάρλινγκ. Δεν έγινε αντικατάσταση της επίλυσης διαφορών κράτους-κράτους ε, από το σύστημα επενδυτικών δικαστήριων στην ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και εμείς έχουμε ένα σύστημα ε, επίλυση κράτο κράτους-κράτους με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ με διαφορετικό βαθμό εφαρμογής, αλλά και στους κανόνες προστασίας επενδυτή μπορούμε να έχουμε κάποιους κανόνες επίλυσης διαφορών κράτους-κράτους. Μερικές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες δεν έχουν ε, όλους τους κανονισμούς αυτούς, όλους τους μηχανισμούς αυτούς. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είναι διαφορετικό το πρίσμα, διαφορετική προοπτική. Θα πρέπει να έχουμε ένα πιο προβλέψιμο, σταθερό σύστημα δικαστικό. Και αυτό κάνει ο ΠΟΕ για τις ε, διαφορές μεταξύ κρατών. Και αυτή είναι η καινοτομία ε, σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή. Να περάσουμε ε, προοδευτικά σε ένα σύστημα που θα είναι ιονίδικαστικό. δικαστικό. Βέβαια έχουμε και άλλα διεθνή σώματα για τις διαφορές μεταξύ κρατών που ε, έχουν τη δικαιοδοσία για τα θέματα αυτά. Δεν είναι βέβαια το ΠΟΕ, εδώ το αρμόδιο όργανο. Και γι' αυτό είμαστε σε τελική ανάλυση υπέρ και έτσι απαντήσω, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εγκαταλείψει το θέμα της πολυμέρειας, ούτε για τους ουσιαστικούς κανόνες, ούτε για την επίλυση των διαφορών. Σαφώς είμαστε υπέρμαχοι αυτό, αυτής της πολυμέρειας. Και από τις 1500 συμφωνίες που έχουμε είχαμε ε, πολύ λιγότερες ε, ευρωπαϊκές που τις αντικαθιστούν, αλλά δεν εγκαταλείψαμε το θέμα της πολυμέρειας, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν μπορούμε να μετακινηθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί θα πρέπει και οι άλλοι να συμφωνήσουν μαζί μας. Και το θέμα είναι τι στρατηγική έχουμε για όλα αυτά θα επανέλθω αργότερα στο θέμα της στρατηγικής. Με ρωτήσατε αν η λογική έχει αλλάξει για τα τοπικά δικαστήρια, τακτική δικαιοσύνη. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν θέλουμε να γίνει καμία αντικατάσταση. Τώρα για το θέμα της Κίνας. Το τι κάνουμε με την Κίνα θα κρίνει και το τι θα κάνουμε και με τη Σιγκαπούρη και άλλες χώρες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Εδώ θα ήθελα να είμαι σαφής. Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε ε, συμφωνήσει στο TTIP είναι ένα ε, σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων όχι μόνο για το TTIP και για άλλες συμφωνίες. Οπότε τα βασικά στοιχεία αυτού του συστήματος θα τα υποβάλουμε και στους άλλους εταίρους μας προς διαπραγμάτευση. Και από την άποψη αυτή έχουμε την προσέγγιση ενός καθορισμένου συστήματος διατησίας και καταθέσαμε τα βασικά στοιχεία και στην Κίνα. Και το προηγούμενο κείμενο έχει πλέον ε, ξεπεραστεί. Και δεν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση του παλιού συστήματος με την Κίνα. Ε, βέβαια, δεν συμφωνούν όλοι 100% μαζί μας. Η πρόταση για το TTIP σίγουρα διαφέρει και η κατάσταση διαφέρει από τη συμφωνία με τον Καναδά. Εκεί έχουμε πλήρω διαμορφωμένο κείμενο. Ε, για τη Σιγκαπούρη δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στις συζητήσεις, αλλά με τον Καναδά έχουμε όχι ένα προς ένα, αλλά σίγουρα ένα πυρήνα των νέων προτάσεων και στη συμφωνία με τον Καναδά. Επίσης έχουμε επαφή με τους συναδέλφους ε, στη Σιγκαπούρη και τους καλέσαμε σε συζητήσεις. Και η αντίδραση που ίσως ε, παρατηρήσατε ε, μετά από τα σχόλια που είπε η κυρία Ροντρίσκη Σπινιέρο προς το παρόν η Σιγκαπούρη απλώς θέτει ερωτήσεις, θέτουν πολλές ερωτήσεις. Και εγώ πιστεύω ότι Έχουμε προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσεις. Η, Συγκαπούρη η Σιγκαπούρη θεωρεί ότι δεν έχει γίνει κύρωση της ε, ε και της ε, προσφυγής που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την καναδική εμπειρία που είχαμε, την εφαρμόσαμε και είπαμε ότι δεν έχει νόημα να αρχίσουμε αναδιαπραγμάτευση άρνητων συμφωνιών. Απλώς με προσοχή ενημερώσαμε για τις πολιτικές. Και καλό ήταν που είχατε άμεση επαφή με τους ομολόγους στη Σιγκαπούρη για να τους δώσετε μια ε, γεύση για το τι σημαίνει πολιτική και ποια είναι η βασική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ε, στείλαμε πρόσκληση και εξακολουθεί να είναι έγκυρη και προς ε, τους ομολόγους μας στη Σιγκαπούρη. Και θα επανέλθουμε στις συζητήσεις. Αλλιώς, ε, αν δεν εκδηλώσουν επιθυμία να προχωρήσουμε στο διάλογο, θα κολλήσουμε. Επίσης, έχουμε ένα σαφές σχέδιο για το θέμα της στρατηγικής ε, για την πολυμέρεια. Και για πολλά χρόνια είχαμε δραστηριοποιηθεί στον ΠΟΕ και μέχρι την υπολική διάσκεψη του Κανκούν ε, που βγήκε από, ε, από το πρόγραμμα της Δόχα, γιατί πιστεύαμε ε, ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι σωστή. Η εναρμόνιση, τουλάχιστον οι σφαιρικοί κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις, είναι οι δύο όψεις του ίδιου Και το ισχύο σύστημα για τις επενδύσεις, αν θέλαμε κάποιους κοινούς κανόνες στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καλό θα ήταν αυτοί να αποφασιστούν πολυμερώς. Δυστυχώς ε, δεν είναι πολλοί ούτε στον ΠΟΕ ούτε αλλού που συμφωνούν μαζί μας υπέρ της πολυμέρειας. Βέβαια δεν έχει λήξει το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και στον ΠΟΕ και αλλού στο μέλλον. Πάντως πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε και άλλες μόρφες, να έχουμε σε μερικά θέματα πολυμερή ε, προσέγγιση, στον ενεργειακό χάρτη για παράδειγμα. Και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε συζήτηση σε ένα πολυμερές δικαστήριο, ίσως αρκεί να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο με ένα συγκεκριμένο ορισμένο αριθμό χωρών. Δεν χρειάζεται να προσυπογράψουν όλες οι χώρες του κόσμου. Και να οδεύσουμε προς ένα πολυμερές δικαστήριο κάτι που θα διαμορφώσει ένα πιο ενοποιημένο ομοιόμορφο σύστημα, ώστε όλο και περισσότερες χώρες να το εστερνίζονται, εγκαταλείποντας σταδιακά τις, διαμερες, τις διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι το σενάριο που θέλουμε να αναπτύξουμε και στο μέλλον. Και έχουμε συζήτηση με πολλές χώρες και προσπαθούμε να τις βολιδοσκοπήσουμε για να δούμε αν ενδιαφέρονται. Πάντω, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζομαι 160 χώρε να προσυπογράψουν ένα τέτοιο σύστημα πολυμερέ για όλε οι χώρε του ΠΟΕ. Στόχο μα είναι ένα πλέγμα πολυμερών συμφωνιών για τα βασικά συστήματα προστασία των επενδύσεων και επίση για τι επιλύσει διαφορών θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα. Αυτό είναι η πρώτη μα προτεραιότητα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα περάσω στα θέματα και τις ερωτήσεις κυρίας Κέλλερ. Μας είπε αν ε, μετανιώσαμε που δεν ε, περιλάβαμε και τη ρήτρα της εκπνοής, στο sunset close. Ε, ό,τι έγινε έγινε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην κατάσταση. δεν μπορώ φυσικά εδώ να μιλήσω στο όνομα των κρατών μελών. Το είδαμε στο TTIP, το είδαμε στην συμφωνία με τον Καναδά και στη συμφωνία με το Βιετνάμ, ότι είχαμε υποστήριξη των κρατών μελών και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Τώρα, για τον Καναδά θα πρέπει να δούμε το θέμα. Προσπαθούμε ε, νομικά να να λύσουμε το θέμα, περιμένοντα την απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν ληφθεί η απόφαση, θα πρέπει να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Για να δούμε αν στο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων έχει μείνει ένα τμήμα αρμοδιοτήτων που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Αλλά αυτό ακόμη μένει ανοιχτό. Και τέλος, ε, ερωτήσεις του Πρόεδρου του κ. Λάγκεν. Τρεις ερωτήσεις υποβάλλατε κύριε Πρόεδρε, που επίσης αφορούν αυτά που είπε και ο κύριος Ζαντό. Εμείς δεν είπαμε ότι υπήρχε άμεση σχέση μεταξύ της ύπαρξη κανόνων προστασία επενδυτών και της αύξησης του όγκου των επενδύσεων. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν έρευνες, άλλοι λένε το μακρύ τους και άλλοι το κοντό τους, άλλοι λένε ότι ε, επηρεάζει θετικά, άλλοι όχι. Η απάντηση είναι ότι βοηθάει ένα πλέγμα κανόνων προστασίας των επενδύσεων. Γιατί αν πηγαίνει κανείς σε μια επικίνδυνη χώρα, φυσικά θα έχει προτιμήσει να έχει εμβολιαστεί για να μην προσβληθεί από μια αρρώστια. Όσο πιο ασφαλής θα είναι κανείς για να κάνει επενδύσεις, ε, τόσο πιο φθηνές είναι και ασφάλεις που θα πρέπει να πληρώσει, μειώνονται τα ασφάλιστρα όταν η χώρα είναι ασφαλής. Όταν δεν έχουμε αποδείξεις ότι μια χώρα είναι ασφαλής και μπορεί να μας να εξασφαλίσει τη συμφέροντά μα, δεν βοηθά κάτι τέτοιο τι επενδύσει. Γι' αυτό θέλουμε σαφή μηνύματα προ του επενδυτέ ότι τη χάνουν προστασία. Και οι εταιρείε και οι επενδυτέ είναι αυτέ που ξοδεύουν χρήματα, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και είναι συμφέρον του να έχουν ασφαλεί ε, ε, και προβλέψιμους κανόνες και ασφάλεια δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Για παράδειγμα, το επενδυτικό κλίμα, το επενδυτικό περιβάλλον επηρεάζεται από θέματα φορολογικά. Για παράδειγμα, άλλη παγκόσμια πρόκληση. Το φορολογικό σύστημα επηρεάζει τις επενδύσεις. Ε, το επίπεδο τη παιδεία και αυτό ε, διαδραματίζει ρόλο. Γιατί τις μεγαλύτερες κινδύνους αναλαμβάνουν οι επενδυτές στις μεγάλες αγορές φυσικά και όχι στις μικρές. Αυτό εξαρτάται και από το μέγεθος των οικονομικών δραστηριοτήτων και το, το κέρδος που αναμένεται. Επίσης, προσπαθούμε να αποφύγουμε ουσιώδεις διαφορές. Επισημένοντας ότι υπάρχουν κάποια κεντρικά σημεία στην προσέγγιση. Το δικαίωμα του νομοθετήν, αυτό είναι κεντρικό σημείο κέριο ή ποιος είναι αρμόδιος, ε, ε, ποιος έχει τη δικαιοδοσία, ποιο δικαστήριο ή άλλος φορέας. Θέλουμε ένα, μια πιο ομοιόμορφη και νομολογία. Και το βασικό μας μήνυμα σε όλες τις ε, συμφωνίες αυτό είναι, ότι υπάρχουν κάποια κεντρικά σημεία που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Αυτά προσπάθησα να απαντήσω. Θα πρέπει να περιμένουμε και τη δικαστική απόφαση για να δούμε τις συνέπειες και θα σας ενημερώσω στο μέλλον ανάλογα με την πορεία. Πρόεδρο Λάγκε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητεί κανεί άλλο τον λόγο. Α, α ναι, ναι, ναι, ναι, α, μάλιστα. Είδα κάποιον. Ε, από τη δική μου τώρα όμως πλευρά, να ξαναρωτήσω, υπενθυμίζοντας πρώτα την ερώτηση της κυρίας Κέλλερ σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή. Δεν είναι μόνο το θέμα δεν είναι μόνο αν θα κριθεί ως μικτός τομέας, αλλά όπως έγινε και στη συμφωνία με την Νότια Κορέα για ορισμένα τμήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, αν θα εξαιρεθούν από την προσωρινή εφαρμογή ορισμένα τμήματα δηλαδή όπως αυτά. Μήπως μπορείτε να επεκταθείτε λίγο και σε αυτό. Και δεύτερο, υπάρχουν και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ συμφωνίας Βιετνάμ, ΣΕΤΑ και ΤΤΙΠ. Η ρήτρα, η umbrella clause στη συμφωνία TTIP υπάρχει, όχι στις άλλες. Είναι ουσιαστικό όμως το ερώτημα αυτό. Όμως, η κύριοι Σόλτς και η Αρίκη νομίζω. Μία πρόσθετη ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Υποχρεώσεις του επενδυτού. Έχουμε δικαιώματα των επενδυτών. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τις υποχρώσεις των επενδυτών μέσα στο σύστημα αυτό και ιδίω σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που μπαίνουν και σε άλλες συμφωνίες και όπου στοχεύουμε στο θέμα αυτό εκεί. Δεν θέτω θέμα των εγγράφων του Παναμά αυτή την είδηση που έσκασε σαν βόμβα σήμερα. Και εγώ θα πλειοδοτήσω σε αυτό το θέμα της ε, προσωρινής το Μιλούμε για την συμφωνία ΣΕΤΑ. Έχουμε ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις και εκεί διευκρινίζεται ότι εάν υπάρχει μια ισχύς προσωρινή της συμφωνίας τότε εκείνο το τμήμα που αφορά το ICS μπορεί να το επικληθεί μια επιχείρηση, να το, επικληθεί, να το επικαλεστεί μάλλον μια επιχείρηση για μια μεικτή συμφωνία εκεί που η σχετική χώρα έχει απορρίψει την σχετική συμφωνία. Δηλαδή ότι έτσι θεσπίζεται ένα παράλογο σύστημα. Ε, καθίστε και σκεφτείτε πώς οι Ευρωπαίοι πρόκειται αυτό να το εισπράξουν. δηλαδή με αυτή τη συμφωνία, ακόμα και αν πει όχι ε, κάποιο κράτος για μια συμφωνία, για τη συμφωνία ΣΕΤΑ, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιος, ας πούμε οι κάτω χώρες λένε όχι στη συμφωνία ΣΕΤΑ. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δίνουν το πράσινο φως. Οπότε υπάρχει μια προσωρινή ισχύ της ΕΤΑ. Οπότε θα μπορούσε επί τρία χρόνια ε, να ανασυρθεί στα δικαστήρια η Ολλανδία από τις επιχειρήσεις ε, επί τη βάση της συμφωνίας. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Άλλη παρατήρηση. Αυτό μας και εμάς ως περισσότερο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμάς ως ΙΝΤΑ, διότι χρειάζεται να μας επιβεβαιώσετε απεβεβαιώστε γιατί τονίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του συστήματος ISDS και της ποσότητας των επενδύσεων. Γιατί είναι τελείως παράλογο να θέλουμε τώρα να αλλάξουμε το νομικό πλέγμα υπέρ των επιχειρήσεων. Χωρίς όμως να υπάρχει κανένα δείγμα ότι αυτό θα φέρει περισσότερες επενδύσεις. Αυτό αλλάζει εκ βάθρων το νομικό πλέγμα που διέπει την κοινωνία μας χώρες, τι να μας αποδίδει κάτι. Άρα το μόνο το οποίο μας λένε είναι ότι η διαδικασία ISDS δεν είναι κάτι το κακό για τις ε, επενδύσεις. Wow, έχω να Γιατί θα πρέπει επομένω να σας πω ότι καμιά φορά πάμε για μια τόσο εκβάθρον αλλαγή, χωρίς να έχουμε κανένα είδους επιχείρημα ότι αυτό θα βοηθήσει τις επενδύσεις. Yes, thank you again. I think... Ο εκπρόσωπος Επιτροπής, ευχαριστώ και πάλι. Πρώτη σας ερώτηση για την προσωρινή εφαρμογή. Εν τέλει νομίζω αυτό θα χρειαστεί περισσότερη πολιτικού χαρακτήρου συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε πουθενά τώρα εδώ, γιατί ταυτόχρονα προβάλλουμε επιχειρήματα και ενώπιον του δικαστηρίου, με την έννοια ότι πρόκειται για ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες μέλη δεν συμφωνούν σε ορισμένες πτυχές που έχουν σχέση με την προσωρινή εφαρμογή και ίσως να μην συμφωνήσει ούτε και το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, ένα πρώτο βήμα θα είναι η... το σχέδιο αποφάσεως της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ακόμα όμως δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση, δηλαδή τι θα μπει στο σχέδιο αποφάσεως για το Συμβούλιο ως περιεχόμενο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα εδώ που θέσατε εσείς κύριε Πρόεδρε για την umbrella clause, δηλαδή το λεξιβροχείο και εκεί έχουμε λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ερώτηση ή μάλλον η απάντηση επ' αυτού είναι ότι η πολιτική της Επιτροπής επ' αυτού είναι υπέρ όχι μιας παλαιού είδου umbrella clause, αλλά μια, μια πολύ συγκεκριμένη και σωστά σχεδιασμένη umbrella clause για να προσφέρει πολύ συγκεκριμένα κίνητρα για τις επενδύσεις, εφόσον δηλαδή έρχονται επενδυτές και υλοποιούν επενδύσεις σε βάση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που έχουν γίνει απέναντί τους. Για να είμαι ειλικρινής, οι Καναδοί και άλλοι έχουν μια πολιτική αλλά και νομικές παραδόσεις και εκεί βρίσκονται οι διαφορές μεταξύ Καναδά και Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έχει πολλές ε, συμφωνίες με umbrella clause, το ίδιο και η Σιγκαπούρη. Από όσο ξέρω ο Καναδάς όχι. Και εκεί οι συμβασμοί που έχουμε, στους οποίους έχουμε καταλήξει είναι διαφορετικοί. Δεν λέω ότι όλα θα είναι απολύτως ισοδύναμα ένα προς ένα, είναι ένα ιδιαίτερο σημείο όπου νομίζουμε ότι οι κανόνες προστασίας που έχουμε διαπραγματευτεί σε ορισμένες συμφωνίες στην ουσία προσφέρουν θεμένη αξία. Έστω και αν αυτό δεν ίσχυε για κάθε μία συμφωνία στο παρελθόν. Για το ερώτημα Σόλτς για τις υποχρώσεις των επενδυτών. Προφανώς οι συζητήσεις μας εδώ έχουν θίξει και το θέμα αυτό και είμαστε κάτι επανάληψη Οφείλω να επαναλάβω ότι κάθε κυρίαρχος χώρα μπορεί να επιβάλλει την ε, δική της νομοθεσία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν υποχρώσεις οι επενδυτές. Έχουν πολλές υποχρώσεις και στην Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια το πολιτικό επιχείρημα εδώ και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και σε επενδυτικές συμφωνίες, δηλαδή να προσπαθήσουμε να πιέσουμε υπέρ μιας σύμφωνης με τη διοντολογία ε, συμπεριφοράς και σύμφωνης με την ομοθεσία όπως αυτή ε, θεσπίζεται από την χώρα υποδοχής των επενδύσεων. Γι' αυτό και έχουμε προτάσεις ε, βιώσιμης, βιώσιμης αναπτύξεως και με τη Μιανμάρ και με την Κίνα και γι' αυτό και προωθούμε θέματα εταιρικής ευθύνης Λέτε εσείς ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως ένας νομικά δεσμευτικός κανόνας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να επιβληθεί μέσω διεθνών συμβάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εάν δηλαδή η χώρα μέλος με την οποία διαπραγματευόμαστε δεν τα συμπεριλάβει στην πολιτική της ως εκ του νόμου απορρέωσες υποχρεώσεις. Προσπαθούμε πάντως και μάλιστα με κάποια σχετική επιτυχία να διασφαλίσουμε ώστε το όλο αυτό θέμα της δεοντολογικής συμπεριφοράς και της βιώσιμης αναπτύξεως να είναι τμήμα των διαπραγματεύσεών μας. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι δεν είναι σημαντικό. Το είναι σημαντικό είναι εδώ και 10-15 χρόνια και του δικού μα επενδυτέ. Για τον κύριο Ζαντό. Θέλω να επανέλθω. Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς πράγματι τη σχέση αιτίου και αιτιατού όταν κάποιοι επενδύουν. Είναι ευκολότερο να δει κανείς καμιά φορά ότι η παραμονή του επενδυτού, της επενδύσεως δηλαδή, οφείλεται στο ότι υπάρχει σύστημα προστασίας. Μιλούμε συχνά τώρα για ένα διεθνές κεφάλαιο το οποίο είναι εντελώ αδέσμευτο και, και, κινείται πάρα πολύ ταχαίω από χώρα σε χώρα. Δεν λέω ότι αυτό επιφέρει κάποια διαφορά. Υπάρχουν μελέτες που λένε ναι και άλλες δεν τα λένε τόσο ξεκάθαρα. Είναι μια πολυσχηδή στην πραγματικότητα συζήτηση αυτή και ίσως κάποια στιγμή μπορούν να εξαχθούν κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Πάντως για την ώρα θεωρούμε ότι ενέχει μεγάλη αξία η ύπαρξη κανόνων. ιδίω αν δούμε και κάποια πρόσφατα παραδείγματα όπου χρησιμοποίησαμε τις διατάξεις αυτών των συμφωνιών σε ορισμένες περιπτώσεις όπου εν τέλει οι Ευρωπαίοι επενδυτές ήταν πολύ ικανοποιημένοι που μπόρεσαν να αποφύγουν μεγαλύτερες ζημίες ε, από τις επενδύσεις που δεν είχαν πάει καλά. Αρκούμε σε αυτά. Ο κ. Ντάουτμοθ. Συγγνώμη, καθυστέρησα γιατί άρχισε το τρένο μου. Και ίσως, ε, ίσως ε, αυτό που θα πω το καλύψατε ήδη μερικός ή ολικός, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να το τονίσω. Έγραψα ένα φυλάδιο αρκετά πολυσέλιδο Είχα αρκετή εμπειρία στην Επιτροπή Τρέιντ και ευχαριστώ θερμά τους ε, συναδέλφους, τον κύριο, τον στόρινο μας πρόεδρο Λάγκε, τον πρώην πρόεδρο ε, Μορέρα. Ε, το μισό φυλάδι αφιερώνεται στο εμπόριο και δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να εντρυφήσω σε άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις και σε ποιο βαθμό καλύπτονται αυτές από τη συνθήκη της Λισαβόνας και επίσης κυρίως πώς οι άμεσες και μια και άμεσα αλλοδαπές επενδύσεις ε, είναι τώρα αρμοδιότητα, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Δεν βρήκα τίποτα, παρόλο που έψαξα α, και αυτό δεν ασχολήθηκα. Ε, ή εν μέρει δεν ασχολήθηκα επειδή είναι περίπλοκο το θέμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς το ζήτημα το πώς άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις ε, ως αρμοδιότητα κοινοτική θα, εφαρμοστούν, θα εφαρμοστεί αυτή η αρμοδιότητα εμπράκτος. Γιατί εμείς προβληματιζόμαστε. Και έχω κουράσει τον αδέρφος γιατί το έχω δηλώσει επανειλημμένος, ίσως και υπερβολικά πολλές φορές. Ανησυχούμε λοιπόν και προβληματιζόμαστε για το τις συνέπειες που θα έχει αυτή υπερβολική ροπή, κρίμα που φεύγει ο κύριο Ζέντο, που είναι υπέρμαχος αυτού του θέματος, τις τάσεις της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλών κομμάτων να συμπεριλαμβάνουν σε εμπορικές συμφωνίες μία σειρά ε, ρητρών και πολιτικά θέματα που δεν έχουν καμία σχέση ή ε, ελάχιστη σχέση έχουν με το εμπόριο. Οπότε, η ερώτηση είναι η εξή. Πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο και με τις άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις. Και αν ε, εσείς το θέλετε, το προτιμάτε, είναι στόχος πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι τέτοιο. Και αν δεν έχετε καταλάβει την ερώτηση, πολύ ευχαρίστω να τη διευκρινίσω. Τελευταία ερώτηση. Καμία από τις δραστηριότητε που συζητούμε και που εξετάζουμε εμεί δεν γίνεται εν γενό και θέλω να σα πω ότι απλά φιλοσοφική ούτω ή δεν σχετίζονται όλα με όλα. Επομένω, θα πρέπει να κάνετε και να σκεφτείτε ε, αυτό που εσεί αποκαλέσατε ε, άσχετε πολιτικέ δεν είναι άσχετε, αφορούν πάρα πολλού. Και νομίζω ότι μπορούμε να εξετάσουμε τι συνάδει, όχι πως κάποια συμφωνία. Και αυτό το κάνουμε σε μια ολόκληρη χρονική διαδρομή. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με ε, τις συμφωνίες, τι γίνεται με τις επενδύσεις. Προσπαθούμε να δούμε τι είδους ρύθμιση είναι η επιθυμητή. Διερευνούμε τι διαπραγματεύσει. Να, όπως ε, και στι διαπραγματεύσει με την ε, Κίνα προσπαθήσαμε και να εντάξουμε και κάποιε ε, κάποιε κάποιες διατάξεις για το περιβάλλον και για τι εργασιακέ σχέσει. Βέβαια αυτό σχετίζεται και με το θέμα του ανταγωνισμού στις επενδύσεις. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο. Είμαι σίγουρο ότι θα είμαστε σε επαφή για την ε, επενδυτική πολιτική και για τις ε, εν λόγω συνθήκες, αλλά και γενικότερα μια που η σημασία της ε, πολιτικής, ε, το σύστημα ICS, ο ενεργειακός χάρτης, όλα αυτά απαιτούν τη εξέταση να δούμε τι γίνεται με τις διμερείς συμφωνίες και ελπίζουμε πριν το 2020 να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθειά μας και να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε σας ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου θέμα, στο 12. Πού είναι τα διάφορα, δεν έχουμε τίποτα. 13. Προσεγγή συνεδριάσει. 20 και 21 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Και η προσκευαστική συνάντηση θα αρχίσει εδώ σε 5 λεπτά και κλεισμένο το θυρών για αυτό το, τον τριμήρη διάλογο